Buenas tardes. Empezamos la reunión. I will speak in Spanish. Bueno, damos aprobado el orden del día, si no hay ninguna observación, y el acta de las reuniones del 10 y el... Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Πρώτα έχουμε τα πρακτικά των οργών συνεδριάσεων που μπορούμε να εγκρίνουμε. Να περάσουμε τώρα στην έκθεση της ε, Επιτροπής του 2016 ε, για την Τουρκία. Πρόκειται για την δεύτερη εξέταση αυτής της ε, έκθεσης. Η Τουρκία έχει περάσει από μια ταραχώδη περίοδο μετά την απόπειρα πραξικοπήματος τον περασμένο Ιούλιο. Είχαμε το δημοψήφισμα τον Απρίλιο με τη συνταγματική μεταρρύθμιση όπου η συνθήκη της Βενετίας έχει αναφέρει σημαντικές ε, επιφυλάξει. Θέλουμε να συνεχίσουμε την παρακολούθηση τη κατάσταση στην Τουρκία. Βεβαίω, ε, μεταξύ εξακολουθεί να ισχύει η κατάσταση τη ανάγκη, δεν έχει αρθεί. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Σταγιάννη, από κοινού με τον Ζαν Κλοντ και τον Ντόναλτ Τάσκ, συνάντησαν τον πρόεδρο Ερντογάν ε, πριν από ένα μήνα και η έκθεση ΑΦΕΤ έρχεται να συνεισφέρει στην συζήτηση αυτή που γίνεται για τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωσης Τουρκίας. Να πω ότι μια αντιπροσωπεία τη Κομισιόν θα επισκεφθεί την Άγκυρα μαζί με την Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πιθανών. Βεβαίω δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πότε θα συμβεί αυτό. Πριν δώσω το λόγο ε, στην, επίτρο, στην ε, εισηγήτρια, συγγνώμη, την Κάτι Πύρη, να σα πω ότι η, ψηφοφορία επί τη έκθεση θα γίνει αύριο το πρωί στι 9. Η Κάτι Πύρη έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους και συζητητές, τη γραμματεία και βέβαια ε, όλο το προσωπικό που κάθε μέρα ε, δουλεύει επί ώρες, επί ημέρες ε, επί της έκθεσης αυτής. Ξέρουμε όλοι σε αυτόν τον νίκο τον εξετάζουμε τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Υπάρχουν πολλές απόψεις για την Τουρκία, αλλά το καλό είναι ότι δεν διχαζόμαστε όπως γίνεται στο Συμβούλιο. Ε, έτσι σήμερα παρότι έχουμε τις διαφορές μας χαίρομαι που όλες οι μεγάλες πολιτικές ομάδες μπορούν να συμφωνήσουν ε, επί της γενικής γραμμής 25 συμβαστικές προτάσεις είχαν υποβληθεί πάνω από 300 τροπολογίες είναι σαφής όμως η γραμμή που ακολουθούμε η δική μας αξιολόγηση και αυτό είναι ομόφωνο ε, είναι ότι το πακέτο που υπευλήθη προς δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια της Κοπεχάγης. Δεν συνάδει. Έτσι λοιπόν το κοινοβούλιο αυτό ζητεί από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον αυτό το συνταγματικό πακέτο εφαρμοστεί θα πρέπει να ε, διακοπούν οι αλεξιακές διαπραγματεύσεις. Εμείς έχουμε μια κοινή θέση και στρατηγική για την Τουρκία ω όργανο είμαστε οι μόνοι, διότι το να μην παίρνει κανεί θέση ή απλώ ο καθένα λέει τη δική του προσωπική θέση δεν οδηγεί σε μια ισχυρή δήλωση. Έτσι λοιπόν, όπω και τον Νοέμβριο, όταν αυτό το κοινοβούλιο με την εξαίρεση 37 μελών μόλι, όλοι λοιπόν υποστηρίξαμε να παγώσουν οι συζητήσει ε, οι ενταξιακέ. Είμαστε και πάλι λοιπόν ενωμένοι σήμερα. Θέλουμε ένα σαφέ μήνυμα αυτή την εβδομάδα ε, θα συνέλθουν και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το δικό μας μήνυμα είναι ενιαίο. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για τη συζήτηση στην Τουρκία εδώ. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ε, σε ό,τι αφορά το ότι δεν υπάρχει βελτίωση. Ένας Αμερικανός δικαστής ε, στην Τουρκία έχει κραδικαστεί για 7 χρόνια. Ένας ένα τρέχο αντιπολίτευση ε, είναι στην φυλακή 25 χρόνια. Σήμερα ε, λαμβάνει χώρα και αυτέ τι μέρε μάλλον λαμβάνει μια μεγάλη πορεία από την Άγκυρα στην Ισταμπούλ οργανωμένη από την αντιπολίτευση ε, με σύνθημα τη δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν και εμεί να στείλουμε ένα μήνυμα προ τον τουρκικό λαό ότι εμεί είμαστε στο, πλάι αυτών που παλεύουν για τη δημοκρατία. Αυτά δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσει εν ώψη της ψηφοφορίας αύριο, εγώ είμαι διατεθειμένη να απαντήσω. Πάντω χαίρομαι ιδιαίτερα και είμαι περήφανη που για τρίτη συνεχόμενη φορά οι σκιώδεις συγητές έπαιξαν ένα πολύ επικοδομητικό ρόλο και έτσι μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αύριο λοιπόν θεωρώ ότι θα υπερψηφιστεί κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτή η έκθεση. Μάλιστα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι σκιώδεις συγητές. Πρώτα η κυρία Μανέσκου παρακαλώ. Ευχαριστώ θα μιλήσω στο όνομα της κυρίας Ζόμερ. Ε, καταρχήν συγχαίρει ε, την εισηγήτρια για τη συνεργασία που είχαν. Πέρσι είχαμε φτάσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με το ψήφισμά μας. Ε, δυστυχώς έκτοτε είχαμε δραματικές εξελίξεις. Ε, είχαμε το ναυπροπλασικοπήματος και το δημοψήφισμα. Υπάρχει συνένεση βεβαίως για σε ό,τι φορά την άποψή μα, αλλά είχαμε αρκετέ αρχικέ διαπραγματεύσει για να φτάσουμε σε συμβασμού. Ε, έχουν πάρθει κάποια δραστικά μάτια μετά, μετά την του πλησιοπήματο. Συμφωνούμε όλοι ότι η απόπειτο δημοψήφισμα ε, δεν συναντηθεί με χάγη Κοπεχάγη. Επίση, καταπιέζονται μια σειρά από ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, συμφωνούμε επίσης για την επίσημη διακοπή των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να, να διακοπούν επισήμως εφόσον το συνταγματικό αυτό πακέτο εφαρμοστεί χωρίς να τροποποιηθεί, διότι οι αλλαγές αυτές δεν ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια της Κοπενχάγης, όπως αυτό αναφέρεται ε, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν με μία φωνή για το θέμα αυτό και θα πρέπει βεβαίως να καταδικάσουμε τη δικτατορική συμπεριφορά του Προέδρου ε, Επίσης ό,τι αφορά τα, τα, τα χρήματα που έρχονται από το IPA, IPA ε, κάποιοι θέλουν να τα παγώσουμε αμέσω, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν γιατί ακόμα να αποστέλνουμε χρήματα στην Τουρκία. Ε, εμείς όμως ζητούμε να παγώσουν τα κονδύλια μόλις παγώσουν και οι διαπραγματεύσεις συνταξιακές. Καταρχήν έχουμε καταστήσει, σαφές ότι τα χρήματα τα οποία έχουμε ήδη υποσχεθεί στην Τουρκία θα πρέπει να αποσταλούν απευθεία στην κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, ιδιαίτερα ε, προς τους πρόσφυγες. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφερθούμε ε, στις ε, πολλαπλές προσβολές που ακούστηκαν πριν το δημοψήφισμα υπόθηκε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε είναι ναζί μεταξύ άλλων. Υπάρχει επίσης το θέμα τη Κύπρου που συζητείται έντονα κάθε χρόνο και το είπαμε και στην περσινή έκθεση αυτό. Αναγνωρίζουμε βεβαίω ότι έχει σημειωθεί πρόοδο στι διαπραγματεύσει ε, του πρόσφατου μήνε. Γενικότερα είχαμε καλέ διαπραγματεύσει. Μπορούσαμε να τα βρούμε γύρω από κάποιου συμβασμού και να φτάσουμε σε ένα καλό κείμενο το οποίο ελπίζουμε ε, θα υπερψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία αύριο.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 το κείμενο ήταν πολύ ικανοποιητικέ. Έχουμε καταλήξει σε κάποιε συμβιβαστικέ, ε, τι οποίε σα συστήνω. Ήταν πολύ καλό που προχωρήσαμε ε, έτσι. Αν το δούμε εξωτερικά, ε, θα πρέπει να δείξουμε ότι ναι, δεν ξεχνάμε την Τουρκία λόγω του δημοψηφίσματος και λόγω των εξελίξεων, αλλά θα πρέπει να είμαστε λογικοί, να μπορέσουμε να σταθούμε στο πλευρό της χώρας Να σκεφτούμε δηλαδή τα συμφέροντα του τουρκικού λαού, αλλά να σκεφτούμε και αυτούς που ζουν ας πούμε στην Γερμανία, ε, πολλοί ε, θα επιστρέψουν, θα ήθελαν να επιστρέψουν και εφόσον ε, επιστρέψουν θα πρέπει να επιστρέψουν σε μια χώρα όπου ισχύουν τα δημοκρατικά δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει κύριος, η κυρία Μπάρμαντ που μόλις έφτασε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Χίλντε. Μπήκα τρέχοντα, οπότε ελπίζω να έχουν νόημα τα όσα θα σα πω, γιατί είναι δύσκολο ούτω ή άλλω να καταλήξει κανεί το ποια είναι η καλύτερη λύση για την Τουρκία. Η συγγήτρια και οι σκιώδει εισηγητέ, μετά από μακρέ διαπραγματεύσει, πιστεύω πω έχουν βρει μία βασική γραμμή ε, που καταρχάς θυμίζει το περσινό μας ψήφισμα όπου αυτό το σώμα ήδη ήθελε να συνδέσει με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου με ε, συνέπειες, με, ειδικά μετά από το πραξικόπημα πέρσι, το οποίο δεν είχε συνέπειες. Έπειτα είχαμε και το δημοψήφισμα όσον αφορά τις ε, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Εμείς ε, σαφώς είμαστε με την πλειοψηφία ότι δηλαδή αν αυτό το, το πακέτο υιοθετηθεί όπως έχει, αυτομάτως και δυστυχώς θα έλεγα ότι θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου η Τουρκία δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια της Κοπεχάγης και δηλώνουμε σαφώς ότι αυτή είναι, αυτός είναι ο πυρήνας της εργασίας που έχουμε κάνει και ε, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε να γίνονται σεβαστές ή, ε, τα δικαιώματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για μειονότητες, είτε πρόκειται για διαφορετικούς τρόπους ζωής, είτε πρόκειται για την εξαρτησία του δικαστικού σώματος και εν πάση περιπτώσει εμείς έχουμε εμφανώς τονίσει αυτές τις βασικές αρχές εδώ και χρόνια ως σώμα και σε, από όλες τις πλευρές και υπεράνω των πολιτικών γραμμών, αλλά αυτό που με λυπεί είναι ότι δεν ε, μιλάμε μιλά τόσο ξεκάθαρα και τόσο ανοιχτά η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και γι' αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό εμείς ως εκπρόσωποι των λαών εδώ να είμαστε σαφείς και να τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή. Όλες οι εξελίξεις αυτές στην Τουρκία έχουν πραγματικές συνέπειες και τέλος να πω ότι αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο προέκυψε τακτικά όταν συζητήσαμε, ε, μάλλον κάθε φορά που συζητήσαμε αυτή την έκθεση. Και είναι σημαντικό εμείς και η ομάδα μας και αυτό το σώμα να μην σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την έκθεση ως ένα χαστούκι στο πρόσωπο των όσων στην Τουρκία ανησυχούν επίσης. Αλλά ωστόσο, αν εμείς δεν υπερασπιστούμε αυτές τις αρχές, ποιος θα τις υπερασπιστεί και πώς αυτό θα εξυπηρετήσει ε, αυτούς που υποστηρίζουν την δημιουργία μιας δημοκρατικής Τουρκίας που σέβεται τις ισορροπίες και σέβεται τα θεμέλια του κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό όσοι παρακολουθούν στην Τουρκία και ζητήσαμε μάλιστα και μετάφραση στα τουρκικά της έκθεσης αυτής και έτσι ελπίζω πως θα καταλάβουν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα και ακούμε, ακούμε τις ανησυχίες των πανεπιστημιακών που είναι φυλακισμένοι, των δημοσιογράφων που είναι φυλακισμένοι, των εκπροσώπων της κοινωνία των πολιτών που είναι φυλακισμένοι, αλλά πιστεύουμε ότι δεν έχουμε μεγάλη επιλογή από το να διατυπώσουμε σαφώς τις αρχές τις οποίες εκπροσωπούμε και βεβαίως πρέπει οι υποψήφιες χώρες να τις στηρούν επίσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω ε, ειλικρινά την Κάτι Πύρη, γιατί για ε, τρίτη χρονιά εργάστηκε συλλογικά και ε, έντιμα με όλους τους σκιώδεις εισηγητές, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία και την κατάληξη σε ένα σχέδιο που χωρίς καμιά αμφιβολία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, χωρίς να αποτελεί έκπληξη, θέλω να σταθώ λίγο στο κυπριακό πρόβλημα επειδή κυρίως αναμένονται οι συνομιλίες ξανά στη Γενέβη στις 29 αυτού του μήνα. Και το κάνω γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι το Κοινοβούλιο και θα πρέπει τα μηνύματά μας να εκπέμπονται ασφαλώς και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο για να πω ότι φαίνεται πως και αυτή τη φορά ή αυτή τη φορά στη Γενέβη θα παιχτεί ξανά το μέλλον των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Και δυστυχώς, θα το πω αυτό, η φιλοδοξία, η πολύ μεγάλη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λύση στο κυπριακό πρόβλημα δεν αντανακλάται κατά την άποψη μου μέχρι στιγμής στις προσπάθειες της. Είναι πολύ πιο ψηλή δηλαδή η φιλοδοξία της από το τι προσπάθειες καταβάλει. Ίσως γιατί η Τουρκία στέλνει το μήνυμα ότι το Κυπριακό δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δυστυχώ σήμερα ο κύριο Γιλτιρίμ στην Αθήνα είπε επίση ότι το Κυπριακό θα είναι θέμα των Ηνωμένων Εθνών. Καταλαβαίνετε ότι αυτέ είναι δηλώσει οι οποίε δεν βοηθούν, ενώ ταυτόχρονα οφείλω να πω ότι πολλέ άλλε δηλώσει Τούρκων αξιωματούχων επιμένουν στην θέλησή του για λύση στο Κυπριακό. Άρα αναμένω από συναδέλφου, γιατί όχι, και από πολλού συναδέλφου εδώ, και από εκπροσώπους τη Κομισιόν και του Συμβουλίου, να δράσουν μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί δεν μένουν πολλές μέχρι τις 29, έτσι ώστε να σταλεί το μήνυμα της πίεσης ε, πάνω στην Τουρκία ε, για να υπάρξει τελικά επίλυση στο Κυπριακό. Πολλοί λένε γιατί μόνο πάνω στην Τουρκία. Η απάντηση είναι απλή. Η Τουρκία είναι η κατέχουσα δύναμη κομματιού ε, της Κύπρου και η κύρια αιτία ως εκ τούτου της μη επίλυσης του προβλήματος. Ασφαλώς υπάρχει και πτυχή ελληνοκυπροκεντρική, να το βάλω έτσι, μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά μακάρι να ήταν μόνο αυτή η λύση, θα ήταν μέχρι στιγμής ε, υλοποιημένη. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση, θα πω δύο φράσεις, αφού στην αρχή ε, της παρέμβασής μου, να θυμίσω, είπα πως σαφώς είναι προς σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν ζητήματα που μας απασχολούν, όπως είναι η πρόταση για επικαιροποίηση ε, της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εμείς δεν μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να επικαιροποιηθεί αυτή η σχέση την ώρα που η Τουρκία δεν εφαρμόζει την υφιστάμενη Τελωνιακή Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με όλα τα κράτη-μέλη και δι' με την Κύπρο. Και ένα ε, δεύτερο ζήτημα που μας απασχολεί είναι το θέμα της ελευθεροποίησης τη βίζα που επίσης ε, δεν εφαρμόζεται ή η Τουρκία δεν δείχνει σημάδια εφαρμογής της όσον αφορά την Κύπρο. Με αυτά κλείνω. Ευχαριστώ ξανά την κυρία Πύρη και όλους τους ε, εισηγητές και καλώ ξανά τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλουν με, οποια με οποιαδήποτε δύναμη έχουν προς την κατεύθυνση οι συνομιλίες οι επόμενες στην Κύπρο να είναι οι τελικές και να είναι ε, ε προς την κατάληξη λύσης του κυπριακού προβλήματος. Ευχαριστώ. Gracias. la palabra señor Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούκνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πύρη για τη σκληρή σας δουλειά. Ε, η δική μας και την οποία εκπροσωπώ τώρα, είναι ικανοποιημένη με την συμβαστική 5 που αφορά την, αναστολή των μεταξιακών διαπραγματεύσεων σε περίπτωση που αρχίσει να ισχύει ένα νέο σύνταγμα, αυτό το νέο σύνταγμα ανεφαλαγών. Ωστόσο γνωρίζουμε πως αυτή η ανησυχία όπως η περιγραφή της ε, ισχύουσας κατάστασης στην Τουρκία είναι πολύ απέχει πόρο από την πραγματική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην χώρα, ιδιαίτερα ε, όσον αφορά την, την δικαιολογία, το πρόσχημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, το κίνημα Γκιουλέν, για να φυλακίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ε, μάλιστα, μόλις ε, πήρα μια αναφορά για μια νέα σύλληψη που μόλις έγινε και μάλιστα επισκέφθηκα την κουρδική, την περιοχή της Τουρκίας πριν από λίγους και αφού φύγαμε, πολλοί από τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλήσαμε συνελήφθησαν πιθανότατα επειδή τους μιλήσαμε. Ε, Ε, φοβόμαστε μήπως ε, επιδεινωθεί ακόμη περισσότερη κατάσταση και εκτελεχθεί σε φίλιο πόλεμο. Αυτά και ευχαριστώ. Μάλιστα, περνάμε στους σκιώδες εισηγητές, ε, μάλλον τους τελειώσαμε. Θα σας δώσω από ένα λεπτό γιατί έχουμε και τη Λατινική Αμερική και έρχεται και ο Προεδρεύων ε, του Συμβουλίου για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη στις 4. Ένα λεπτό λοιπόν παρακαλώ. Χριστοφόρου. Είναι ένωση αρχών και αξιών και οφείλουμε όλοι εμεί να τι υπερασπιζόμαστε. Η Τουρκία συνέθλιψε και παραβίασε συλλήβδη κάθε αρχή και αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το χειρότερο και το σημαντικότερο είναι ότι η Τουρκία παραβιάζει αρχέ και αξίε που έχουν να κάνουν με άλλε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζει να προκαλεί και να παραβιάζει τόσο τον εναέριο χώρο όσο και τον θαλάσσιο χώρο τη Κύπρου και τη Ελλάδο, χωρί να υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το σημαντικότερο και το κυριότερο, ενώ συνυπέγραψε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρωτόκολλο της Άγκυρας, δεν το εφαρμόζει. Γι' αυτό είναι πάγια τακτική αλλά και προσβολή προς την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη δεν εφαρμόζει την υφιστάμενη Τελωνιακή Ένωση. Και όταν ακούω αναβάθμιση τη Τελωνιακή Ένωση, όταν δεν εφαρμόζει για μια χώρα μέλο, ήθελα να ξέρω πού είναι η αλληλεγγύη των άλλων χωρών μελών για την Κύπρο, όπου δεν εφαρμόζεται η Τελωνιακή Ένωση. Θέλω να πω για το Κυπριακό ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, ο Νίκο Αναστασιάδη, καταβάλει το άπαν των δυνάμεών του για την επίλυσή του. Όμω, πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση εάν η Τουρκία συνεχίζει να ζητά με θράσο και απροκάλυπτα που παραβιάζει κάθε αρχή οι εγγύσει και η ασφάλεια τη Κύπρου, χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να επαφείται στην Τουρκία. Αυτό προσβάλλει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να απαιτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια να είναι εγγύτρια τη ασφάλεια τη Κυπριακή Ένωση. La Η και οι υπόλοιποι έχουν περιγράψει νομίζω με τον πιο παραστατικό τρόπο την κατάσταση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα σημείο και έχει λεχθεί και από άλλου συναδέλφου. Στην προσπάθεια τη Κομισιόν για να αναβαθμιστεί η τελωνιακή σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Τι σκοπιμότητε εξυπηρετεί πέραν οικονομικών συμφερόντων ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερόντων και τουρκικών οικονομικών συμφερόντων αυτή η πιθανή αναβάθμιση. Τι μήνυμα δίνει στο εσωτερικό τη Τουρκία, τι παιχνίδι παίζεται σε σχέση με τι σχέσει με τον ίδιο τον κύριο Ερτογάν, ο οποίο καθημερινά σκληραίνει τη στάση του. Νομίζω είναι καταστροφική πορεία αυτό που ακολουθείται από πλευρά τη Επιτροπή να προσπαθεί να αναβαθμίσει σχέσει με μια χώρα που δεν σέβεται καμία αρχή. Muchas gracias. Eh, la uh, uh, Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Κάτι και όλους όσοι μπόρεσαν να συμβάλλουν στη σύνταξη της έκθεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο να δώσει ένα ξεκάθαρο και ισχυρό μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα δεν απευθύνεται μόνο προς τον κύριο Ερντογάν, αλλά απευθύνεται κυρίως στον τουρκικό λαό, με τον οποίο ε, αισθανόμαστε αλληλεγγύη. Και εκείνος είναι που χρειάζεται όντως την αλληλεγγύη μας. Ε, επικρίνουμε εντόνως τη δικτατορία του Ερντογάν που όχι μόνο σαφώς παραβιάζει τα κριτήρια της Κοπενχάγης αλλά παραβιάζει και τα δικαιώματα των ανθρώπων και επίσης επιχειρεί να ε, κλείσει το στόμα όλων, ε, φασανιστήρια, δολοφονίες ε, στα κέντρα κράτησης που δεν αναγνωρίζονται ούτε καν από την κυβέρνηση. Την περασμένη μόλις εβδομάδα ο κύριος Εντρογάν έδωσε μια συνέντευξη σε, ένα πορτογαλικό κανάλι τηλεόρασης όπου, μάλιστα κατηγόρησε τους δημοσιογράφους τον δημοσιογράφο, επειδή του απέφθινε την επίκριση ότι θέλει να κάνει τρομοκρατική προπαγάνδα και ότι είναι ε, πραξικοπηματίας ο Πορτογάλος δημοσιογράφος, ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσης με την Τουρκία δεν είναι κάτι το πρόσφατο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι διεξάγονται επί δεκαετίες και καρκινοβατούν συνεχώς χωρίς καμία πρόοδο οφείλαμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η Τουρκία, πώ συμπεριφέρεται, τι στόχου έχει και κυρίω το τι δεν θέλει να κάνει. Παρ' αυτά εμεί εξακολουθούμε να τα χαϊδεύουμε. Παρά το γεγονό ότι οι εκθέσει οι οποίε γίνονται συνήθω κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στροφακομιλίζει και να πιστεύει ότι αν χαϊδεύσει την Τουρκία, αν τη ικανοποιήσει όλε τι απαιτήσει, θα αλλάξει η Τουρκία συμπεριφορά ούτε θα πάψει να απειλεί την Ελλάδα, ούτε θα πάψει να απειλεί την Κύπρο, ούτε θα πάψει να μην αναγνωρίζει την Κύπρο, αλλά παράλληλα θα απαιτεί όλο και περισσότερα. Άρα λοιπόν, μια πραγματιστική πολιτική απέναντι στην Τουρκία λέει ότι πρέπει αυτή να είναι σκληρή. Να διακόψουμε άμεσα τη χρηματοδότηση, γιατί διαφορετικά η Τουρκία θα επιβραδύνει τι διαδικασίε χωρί να επισημειώνεται καμία πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι συγκρίνοντας αυτή την έκθεση με το παρελθόν, ε, η θέση της εισηγήτριας ήταν ακόμα πιο δύσκολη, όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξε σημαντική ανταπόκριση στα θέματα του κειμένου με το τι συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία. Ένα σημείο όμως θέλω να θέσω στην αγαπητή μου Κάτι Πύρη. Θα ήθελα να πάρω μια εξήγηση γιατί η τροπολογία για επιβολή εμπάρκο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις πωλήσει όπλων προς την Τουρκία μετά και την απόφαση της Γερμανίας και της Αυστρίας δεν υιοθετήθηκε στην έκθεση. Εκεί όμως που εκφράζω την απογοήτευσή μου είναι σε ένα γενικότερο επίπεδο που αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Τουρκίας ειδικά προς την δημοκρατία της Κύπρου. Και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το σημείο. Μιλάμε για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είναι ο σεβασμός του, των κανόνων δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι θέμα άποψης. Αυτό αφορά δύο λέξεις και τελειώνω και το θέμα αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης και το θέμα των απειλών στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και επίσης Termine, στο θέμα favor. του κοινοτικού γεχτημένου στα κατεχόμενα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία. σε Ένα πολύ περίπλοκο θέμα που εγώ παρακολουθώ εδώ και αρκετά χρόνια εδώ στο Κοινοβούλιο και μάλιστα μαζί με διάφορους άλλους ευρωβουλευτές. Ε, πιστεύω πως αυτό που μας επιτρέπει αυτή η έκθεση είναι να στείλουμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία και την τουρκική κυβέρνηση όπου λέει σαφώς ότι για το Ευρωκοινοβούλιο τελείωσαν τα ψέματα ε, στη σχέση μας με την Τουρκία, το όσα έγιναν ε, την περασμένη χρονιά και κυρίως ε, η συνταγματική μεταρρύθμιση με σοάδικης εκστρατείας έχει ξεπεράσει οποιοδήποτε όριο που μπορούσαμε εμείς να δεχτούμε για να μπορέσει κάποτε να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Τώρα θα πρέπει από κοινού να σκεφτούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το, το διάβλο επικοινωνίας μέσω της Ελληνική Ένωσης, μέσω ποιου ε, καναλιού θα συνεχίσουμε. Γιατί αυτό ήταν ο τρόπος μας να διαπραγματευτούμε και να, να, να ε, συνεχίζουμε έναν διάλογο. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ποπόσκι. Uh, uh, uh, Σα ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε την ε, προσπάθεια τη εισηγήτριας και των σκιωδών ε, εισηγητών να ε, καλύψουν όλες τις πτυχές των σχέσεων με την Τουρκία. Είμαστε Μάλλον συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράζονται, τις έχουμε εκφράσει και εμείς επανειλημμένως, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάσταση της ελευθερίας έκφρασης του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ανησυχούμε πολύ όσον αφορά την, ε, την, την ελευθερία τύπου και έκφρασης, τα, Επίσης μας ανησυχούν τα όσα καταγγέλει η Διεθνής Αμνηστία ε, και τα όσα συνέβησαν με τον ε, Τούρκο δικαστή του ΟΗΕ η αυθαίρετη, και επίσης μας ανησυχεί η αυθαίρετη εφαρμογή αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Ε, εν γέννη συμφωνούμε με τα απορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν ε, του 2016. Όμως ε, η Τουρκία παραμένει μία από τις πιο κοντιν, τους κοντινούς και σημαντικούς εταίρους. Θέλουμε η Τουρκία να έρθει πιο κοντά στην Ένωση και όχι να απομακρυνθεί από την Ένωση και γι' αυτό και είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την επαφή και αυτό ήταν και το μήνυμα προς τον Τούρκο Πρόεδρο, το οποίο διαβίβασαν οι δύο πρόεδροι Γιούνκερ και Τούσκ στις 25 Μαΐου που αναφέρατε προηγουμένως. Διάφορες ε, ε, συναντήσεις υψηλού επίπεδου έχουν σχεδιαστεί τους επόμενους μήνες. Πρόκειται να ε, σχεδιαστούν για κοινού τομεί συνεργασία όπω η ενέργεια, οι μεταφορέ, η οικονομία, ο ενισχυμένο πολιτικό διάλογο. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μα για τη μετανάστευση μέσω τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες. Στην Τουρκία η συζήτηση για το νέο, την, μάλλον την εντολή για την ανανέωση και τον εξυγχρονισμό της Ελληνικής Ένωσης συνεχίζεται. Τέλος, θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι η δέσμευση μας και οι επαφές θα συνεχιστούν, αλλά ότι βεβαίως θα συμπεριλάβει σε όλα αυτά πολύ στενή παρακολούθηση ε, των, της εφαρμογής των συνταγματικών ε, τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπόφσκη και ευχαριστώ όλους για την ε, κατανόησή σας και για την ταχύτητα. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε και τον Ιούλιο θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Υπήρξαν κάποια ερωτήματα και σχόλια, οπότε αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις. Για παράδειγμα, όταν το ζήτημα αφορά την Τελωνιακή Ένωση, η συμφωνία την οποία έχουμε προσεγγίσει είναι η ίδια την οποία είχαμε προσεγγίσει όταν η ΑΦΕΤ συζητούσε ε, την θέση της ε, σχετικά ε, με την Τελωνιακή Ένωση. Οπότε δεν έχει αλλάξει η θέση μας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η Κυπριακή κυβέρνηση που δεν συμφωνεί με αυτή τη θέση ε, γνωρίζουμε ότι και η Ελλάδα δεν συμφωνεί αυτό. Με αυτό όμω η πλειοψηφία έχει ψηφίσει ε, για αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να αλλάξουμε ε, τη θέση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμω πιστεύουμε ότι έχουμε ε, πάλι μία ισχύ απέναντι στην Τουρκία όσον αφορά την οικονομία. Η οικονομία λοιπόν είναι η, η μόνη δυνατότητα που έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξει η συζήτηση σχετικά με την Ελληνική Ένωση αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό σε περίπτωση που είμαστε βέβαιοι ότι η Τουρκία θα το εφαρμόσει αυτό με όλα τα κράτη-μέλη και τα 28. Όσον αφορά την Κύπρο, ε, συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφος κ. Χατζηγιώργου, ε, χρειαζόμαστε ε, μια επιτυχημένη εξέλιξη των συζητήσεων που θα γίνουν τέλη του μηνός, θα αποφέρουν ένα ευθέο αποτέλεσμα ε, και ε, το οποίο θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την ε, δημοκρατία της Κύπρου. Δεν ρίχνουμε κατηγορίες, ακόμα βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις, δεν λέμε ακόμα ποιος φταίει. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε την διαδικασία και γι' αυτό το λόγο δεν θα δοκιμάσουμε κάτι το οποίο δεν είχε αποτελέσματα πέρσι. Ε, τώρα τα υπόλοιπα ε, σχόλια άκουσα ότι στις διαπραγματεύσεις ε, με, ε, τους, με τον συνάδελφό σας είχαμε μια πολύ καλή συμφωνία πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Δεν αναγνωρίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, ε, πιο ήρεμη γλώσσα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί όσον αφορά τις ελλείψεις των βουλευτών, των δημοσιογράφων, αλλά και όσον αφορά την κατάσταση στις φυλακές, αλλά και στα νοτιοανατολικά της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο αυστηρή γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο λόγος που δεν χρησιμοποιούμε την έννοια εμφύλιος πόλεμος είναι διότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αναγνωρίζει ε, το ε, ΠΚΚ ως μια τρομοκρατική ανοργάνωση και θα πρέπει λοιπόν ε, να αναγνωρίσουμε ότι εφόσον το αποκαλέσουμε αυτό εμφύλιο πόλεμο τότε είναι σαν να μην ε, φέρει την ευθύνη το ΠΚΚ. Η κατάσταση ναι, είναι ε, τρομακτική. Έχουμε 500 μισό εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους όμως η φράση εμφύλιος πόλεμος έχει μια πολιτική σχέση έχει ένα πολιτικό δίνει μια πολιτικά έννοια την οποία δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε ακόμα σε αυτό το κοινοβούλιο. Το ε, κοινοβούλιο αυτό δεν είναι δικαστής ε, και δεν έχουμε άλλες αποφάσεις σχετικά με το ε, ποιος κρύβεται και ποιος όχι πίσω από το πραξικόπημα και γι' αυτό το λόγο όλες οι τροπολογίες που σχετίζονται με αυτό καταλήξαμε σε μια συμφωνία ότι ακόμα περιμένουμε αποδείξεις όσον αφορά τους ηθήνοντες του πραξικοπήματος. Ε, κύριε Παπαύσκη, όσον αφορά τα σχόλιά σας ε, ε, και στο Κοινοβούλιο εμεί θέλουμε η Τουρκία να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουμε να τους απομακρύνουμε από εμά, όμως νομίζουμε ότι υπάρχουν συνέπειες σε ορισμένες δράσεις και θα πρέπει λοιπόν έχουμε την ευθύνη να διατηρήσουμε την αξιοπιστή μας το πλαίσιο του 2016 είναι δεκάθαρο και, σε περίπτωση, και εφόσον υπάρχουν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφόσον δεν τηρούνται τα κριτήρια της Κοπενχάγης θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις. Σας ευχαριστώ. Βιαζόμαστε για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τους υπόλοιπους εισηγητές. Οπότε περνάμε αμέσως στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η δεύτερη εξέταση της έκθεσης Ευρωπαϊκής, ε, μάλλον πρωτοβουλίας για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική. Ε, εισηγητής είναι ο κύριος Χαβιέρα Λόπες. Ε, έχουν υποβληθεί 258 τροπολογίες από πλευρά των συναδέλφων και στην πρώτη συζήτηση έγινε ε, συζήτηση και με τους κοιόδης συζητητές όπου συζητήθηκαν πολλές συμβιβαστικές. Ο κύριος Λόπες. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ ησυχία καθώς αποχωρείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αρχαία είναι ότι είχαμε μια συζήτηση επί του σχεδίου κειμένου, οπότε θα κάνω μόνο κάποια σχόλια για τις 258 τροπολογίες που έχουν υποβάλει πολλοί από τους και ε, αλλά και διάφοροι άλλοι βουλευτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για την έκθεση. Οι τροπολογίες σε γενικές γραμμές βελτιώνουν το κείμενο, το συμπληρώνουν. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε σε ευρεία συνένεση στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες αναχώρα. Ε, υπάρχουν στοιχεία ε, στα οποία θέλουμε να υπάρξει συμβιβασμός, ε, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε και τη γενικότερη φιλοσοφία του αρχικού κειμένου. Δηλαδή αυτή η έκθεση θέλει να δώσει μια όθηση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής, να τις επικαιροποιήσει. έχουμε το νέο διεθνές ε, περιβάλλον, αν θέλετε, το οποίο αλλάζει κάπως τα πράγματα, το είπαν και οι αυτό και επικεντρωνόμαστε λοιπόν στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ε, τις σχέσεις αυτές ε, και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Προσπαθούμε να έχουμε μια οριζόν, οριζόντια προσέγγιση αλλά και συμμετρική, δηλαδή δεν θέλουμε ε, να κάνουμε μια έκθεση που θα λέμε τι πρέπει να κάνει ο άλλος, ε, θέλουμε πώς να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και πώς μπορούμε χέρι-χέρι να αντιμετωπίσουμε τις ε, παγκόσμιες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η διεθνή κοινότητα. Αναφέρθηκαν κάποια πολύ θετικά στοιχεία στις τροπολογίες αυτές. Ε, να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τις μεγάλες συμφωνίες που είναι υποδιαπραγμάτευση, που είναι στη διαδικασία έγκρισης και αυτό είναι πολύ θετικό. Να γίνεται αναφορά στη διάφορα προβλήματα της περιοχής και αυτό είναι θετικό. Θέλουμε να έχουμε αυτή την οριζόντια προσέγγιση βέβαια όπω είπα. Υπάρχουν και κάποια σχόλια για επιμέρου δυσκολίε που υπάρχουν με κάποιες χώρε. Ε, υπάρχουν διαπραγματεύσει επ' αυτού εδώ, έχουν γίνει στο παρελθόν δηλαδή, οι οποίε αποτελούν σημείο αναφορά, αλλά εντό των επόμενων εβδομάδων ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια ευρεία συνένεση που είναι και ο στόχο μα. Να ευχαριστήσω όλου, ε, ιδιαίτερα τους και ε, για τι προτάσει του. Ευχαριστώ ο Λουίς Δεγκράντες τώρα έχει τον λόγο, παρακαλώ. Όποτε μπορέσετε βεβαίως. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Το τηλέφωνο πάντα χτυπάει την ακατάλληλη στιγμή. Ε, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά η στάση του εισηγητή ε, είναι αξιοπρόσεκτη, ήταν πάντα διαθέσιμος, ήταν συνεργάσιμος ήταν ανοιχτό στο διάλογο. Οι συμβιβασμοί δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά πιστεύω ότι αποτυπώνουν μέχρι στιγμή, μέχρι στιγμή οι νέε διατυπώσει της θέσης μα. Ε, οι τροπολογίε μα έχουν ληφθεί υπόψη. Ε, οι αξίε που θέλαμε εμεί να αποτυπώνονται σε αυτή την έκθεση. Συμφωνούμε με την προσέγγιση του εισηγητή. Δεν θέλουμε εμεί να απαιτούμε δεν έχουμε άλλωστε εμείς ε, την, ε, ε, το δικαίωμα να ζητήσουμε κάτι τέτοιο από τους εταίρους μας. Είναι μια σχέση ισότιμη. Μπορεί να δίνουμε κάποιες συμβουλές, αλλά σε κανένα περίπτωση δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι, διότι δεν μπορούμε να δώσουμε μαθήματα σε κανέναν. Αλλά υπάρχουν κάποιες κοινέ αξίες. Η έκθεση αυτή αναφέρεται σε αυτήν την ε, ένωση των δύο αυτών μεγάλων περιφερειών, δηλαδή Λατινική Αμερική και Ευρώπη, έχουμε κοινά συμφέροντα, ε, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αλληλεγγύη, η ειρήνη, του κράτους δικαίου. Αυτές οι αρχές ε, είναι αρχές αδιαπραγμάτευτες, ε, τις οποίες συμμεριζόμαστε και πρέπει αυτό να είναι καθολικό. Είναι μια ευκαιρία μια στρατηγική εξωτερική πολιτική τη Ένωση, ε, να προχωρήσουμε στον τομέα των ελευθεριών, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ε, γίνονται προσπάθειε τα τελευταία δεκαετία ε, για να υπάρξουν δημόσιε πολιτικέ ε, συμπεριληπτικέ για να προστατευτούν οι πιο ευάλωτε ομάδε, για την αναδιανομή του πλούτου και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό το συμμεριζόμαστε απολύτω. Ε, Βεβαίω δεν πρέπει να υπάρχουν μανιχαϊσμοί, δεν πρέπει να πούμε ότι αυτό το ζητάει μόνο κάποιο. όχι. Το συμμεριζόμαστε όλοι. Έτσι λοιπόν συμφωνούμε και με και τα μέτρα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ε, το, την, καταπολέμηση της διαφθοράς, των λαθροπαρίων ναρκωτικών. Υπάρχουν κάποιες αρχές ε, πολύ σημαντικές να υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τις ε, επενδύσεις, ε, καταπολέμηση της διαφθοράς, αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Είναι σημαντικές αρχές, σημαντικές αξίες που πρέπει να μας ενώνουν. Ε, έτσι ώστε αυτή η σημαντική περιοχή, η φιλική αυτή περιοχή προς εμάς, ε, να συνεισφέρει στην ευημερία ε, των κοινωνιών μας. όλα αυτά αποτυπώνονται αρκετά καλά στην έκθεση. Δεν έχει κλείσει βέβαια ακόμα το κείμενο, αλλά χάρη στο διάλογο έχουμε φτάσει σε, κάποια, σε κάποιες συμβαστικές λύσεις, σε κάποιους συμβασμούς Τέλος, υπάρχει και ανησυχία αυτής της έκθεσης, ε, αυτής της έκθεσης και ε, του Κοινοβουλίου για τη Βενεζουέλα. Εδώ απλώς διαπιστώνουμε ε, την ανησυχία που υπάρχει, διότι, διότι, υπάρχει μια σημαντική επιδείνωση σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, ε, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να μπορέσει να λειτουργήσει, θα πρέπει να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, θα πρέπει να είναι ελεύθερες και διαφανείς οι εκλογικές διαδικασίες. Ε, αυτό φαίνεται και στις συζητήσει ότι υπάρχει η αιμοφωνία από αυτό. Ελπίζω και το θέμα της Κούβας να μπορέσουμε να επιλύσουμε ε, με ένα λογικό τρόπο. Το συζητάμε. Το συζητάμε όλα αυτά. Αυτά, Πρόεδρε, νομίζω ότι αρκεί να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την στάση του ε, και το γεγονό του λάβει υπόψη τη ανάποψή μα. Λοιπόν, επειδή έχουμε στι 4 σημαντική επίσκεψη. Τρία λεπτά να μιλάνε παρακαλώ οι σκιοδεσηγητές. Παρακαλώ επομενο Ναι, σύντομα, η δουλειά του Χαβιέρ είναι πραγματικά εξαιρετικά θετική, είναι πολύ καλή και η στάση του αλλά και η δουλειά του και είμαι βέβαιο ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία, λέει ο κ. Νάρτ. Ευχαριστώ. Μάλιστα, όντω ήσασταν πολύ σύντομο. Θα πρέπει να μιλήσω και εγώ τώρα εκ μέρου τη Γκουε να, καλωσο... να ευχαριστήσω τον Χαβιέρ Λόπεθ και να τον συγχαρώ. Έκανε πολύ καλή δουλειά μπόρεσε έτσι να ικανοποιήσει όλους. Εμείς ήμασταν στην διάθεση βεβαίως του κυρίου ε, εισηγητά, όταν όμως υπάρχουν, ε, υπάρχει ανισορροπία και όταν ε, επιτεθόμαστε σε κάποιες χώρες σχέση με άλλες, τότε και εμείς θα μπορέσουμε προφανώς να υποστηρίξουμε προσπάθειες που θα χαλάσουν την ισορροπία στο κείμενο. Ο κύριος Μπρόκ έχει το λόγο τώρα, παρακαλώ. Όχι. Α, συγγνώμη. Ο κύριος Αλαφράγκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να πω ότι ευχαριστώ τον εισηγητή, το επικοδημητικό του πνεύμα. Όντως αυτό που θέλουμε ε, είναι να φτάσουμε σε μια στρατηγική διαπεριφερειακή ε, σχέση και να την ενισχύσουμε. Να πω ότι αυτό που είπατε για τις τροπολογίες ε, νομίζω ότι για συμφωνίε όπω με τη Βραζιλία και το Μεξικό, με την Αργεντινή, τι μεγάλε χώρε, είναι σημαντικό να υπογραμμίζουμε τη σημασία των προθεσμιών για τι συμφωνίε με το Μερκοσούρ ε, και τη Χιλή και το Μεξικό. Ε, νομίζω ότι αυτό κάνει ο συγητή. Ε, επίση πρέπει να υπογραμμίσουμε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα συνέντευξη ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Και επίση ο νομίζω ότι θα φτάσουμε θα φτάσει σε μια συνένεση, εμεί είμαστε στη διάθεσή του. Εγώ πάντως θα να σα ευχαριστήσω για τι δικέ μου τροπολογίε γιατί ήσασταν εξαιρετικά θετικά διακείμενο. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή πάει πολύ καλά και νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη υποστήριξη από, την, από το Κοινοβούλιο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μιγιαμόν. Ευχαριστώ την τον κύριο Λόπε για το ανοιχτό του πνεύμα και για την ε, ευγένειά του όσον αφορά τι ε, τροπολογίε μα, όχι μόνο των σκιωδών, αλλά και εκείνου που έχουμε έδρανα που, και που ασχολούμαστε με, αυτά τα θέματα. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι και αυτό που είπε ο Λουίς Δεγκράντες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι λατινοαμερικάνικες χώρες θα πρέπει να είναι φυσικοί σύμμαχοι λόγω των πολλαπλών συνδέσμων, συμφερόντων, αξιών και ανθρώπινων δεσμών και της ιστορίας που έχουμε κοινής. Οι τροπολογίες, ε, και μιλώ για τις δικές μου γιατί αυτές γνωρίζω καλύτερα, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Λόπες, ε, τον εισηγητή, να δείξει μία ε, ανοχή όσον αφορά την τροπολογία 145 για κατάργηση. Ε, δεν έχουμε άλλου ομιλητέ, ε, κύριε Λόπε, θέλετε να κλείσετε. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια συνάδελφοι και τα σχόλια των σκιωδών αλλά και των όσων ε, πήραν το λόγο και όντως ήταν επικοδομητικό το πνεύμα όλων των συνεδριάσεων και των, του διαλόγου που κάναμε τις τελευταίες εβδομάδες και να προσθέσουμε και, κάποια πράγματα όπως σωστά είπε ο κύριος Λουίς Δεγκράντες αυτή η έκθεση αυτό που θέλει είναι να ε, προτάξει τις κοινέ αρχές τις κοινέ αξίες, το κοινό θεματολόγιο ε, σε διεθνέ επίπεδο, εκείνα τα θέματα δηλαδή που θα πρέπει από κοινού να μας απασχολήσουν και τρίτον να ε, μιλήσει για τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε αυτές μας τις ήδη ισχυρές σχέσεις. Και σε σχέση με αυτό που σχολιάσατε τώρα, η Λατινική Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμφίβολα είναι καλή, είμαστε καλοί φίλοι. Αυτό που είναι απαραίτητο να είμαστε περισσότερο σύμμαχοι ε, στο διεθνέ προσκήνιο. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας ε, συμμαχία υπέρ ε, των πολυμερών ε, οργάνων, ε, της καταπολέμηση ε, των κλιματικών αλλαγών, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, τη δημοκρατία, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό του Διεθνού θεματολογίου που είναι κοινό και που σήμερα χρειάζεται ισχυρές φωνές και σταθερέ συμμαχίε εντό των μεγάλων πολυμερών οργανισμών, από τον ΟΗΕ μέχρι τον ΠΟΕ και την υπεράσπιση των ανοιχτών κοινωνιών που πλέον ε, δεν βρίσκουν απέχηση σε, σε πρώην ε, ισχυρούς μας συμμάχους. Ενώ με τη Λατινική Αμερική μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες. Και αυτό είναι σημαντικό ε, όσον αφορά την ποιότητα των θεσμών και την ποιότητα των σχέσεων. Σταθερότητα, λοιπόν, και καλή χρηστή διαχείριση. Έχουμε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά στη Λατινική Αμερική από ό,τι στην Ευρώπη, αλλά έχουμε κοινού στόχους. Ε, έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια και για πολλούς και διάφορους λόγους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όμως υπάρχει θέμα με την ασφάλεια στην Λατινική Αμερική όπως και εδώ. Επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαφράγκα που προσφέρει με τη δική του συμβολή και χάρη στη γνώση που έχει ε, όλη της ε, Λατινικής Αμερικής ε, που σίγουρα τα όσα μας προσέφερε θα σε βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την έκθεση αυτή. Λαμβάνοντα υπόψη τι πλειοψηφίε και τι προηγούμενε θέσει του Ευρωκοινοβουλίου, ελπίζουμε πω θα έχουμε μια καλή πλειοψηφία για να μπορέσουμε έτσι να εστιάσουμε στι ε, ε, σχέσει μα. Υπάρχουν κάποια θέματα που είναι περίπλακα στη διαχείρισή τους για, όταν μιλάμε πιο συγκεκριμένα για κάποιες χώρες, ότι θα πρέπει να βρούμε μια κάποια ισορροπία. Ε, και με την Κούβα που στις επόμενες μέρες ε, θα σταθεροποιήσει ε, την σχέση της. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους κοιόδης όλους για την συνεργασία που στόχο είχε να εμπλουτιστεί το κείμενο. Είμαι στη διάθεση όλων ε, για να βρούμε όσο γίνεται μεγαλύτερη συνένεση, ώστε να μπορέσουν ε, και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να σταθούν ε, δίπλα μας στη σχέση μας με τη Λατινική Αμερική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λόπεθ και να θυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιούλιο και εδώ και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Και τώρα διακόπτουμε για να υποδεχτούμε τον Υπουργό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Vamos Ας συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Να καλωσορίσω τον κύριο Σβίζιτς, που είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ο κύριος Ζήτη ε, συνοδεύεται από την πρέσβυρα Τόβες, καλωσορίσατε, και καθώς και από τον Διευθυντή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, τον κύριο Λιβερόβη. Και θέλω να καλωσορίσω δε τους βουλευτές ε, από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη που είναι σήμερα εδώ στο σεμινάριο για την ε, ε, δυνατότητες ε, του εκλογικού κύκλου εδώ στην Ευρωκοινοβούλιο. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Πρόκειται για τη συνέχεια ε, που δίνουμε στην επαφή που είχαμε με τον κύριο Σουρβίκ, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Απρίλιο. Ε, συγγνώμη, τον κύριο Ναρντάκ. θα σας δώσω το λόγο χωρίς άλλη καθυστέρηση. Κύριε Σφίτιτς. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή και χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για άλλη μια φορά για να μιλήσω για την ένταξη της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το να γίνουμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα μου. Θα ήθελα να πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Βοσνίας και της του οποίου προεδρεύω, αφιερώνεται στο να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα οδηγήσουν στην ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση για μας σημαίνει ε, εξυγχρονισμός, σημαίνει εκδημοκρατισμός της χώρας μας. Είναι κάτι που επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις ε, προς όφελος όλων των ε, συμπολιτών μας. Χαίρομαι που οι ευρωπαϊκές αρχές αναγνώρισαν την προσπάθεια που έχει γίνει και ότι αυτό συμπεριλήφθηκε στην έκθεση του 2016. Οι Βοσνία και η Ριζοβαβίνη αναγνωρίζουν επίση ε, τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των θεσμικών τη οργάνων και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να βοηθήσουν τη Βοσνία στον δρόμο προ την Ευρώπη. Όχι μόνο τη Βοσνία, αλλά το σύνολο τη περιοχή. Στη συνάντηση με την ύπατη εκπρόσωπο στα τέλη του περασμένου μήνα στι Βρυξέλλε, ε, στείλαμε ένα πολύ σαφέ μήνυμα. Ε, υπάρχει μια ανοιχτή προοπτική να αποτελέσουμε μέρο τη Ένωση, όχι μόνο εμεί, όλε οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό αναφέρεται και στα συμπεράσματα του τελευταίου Συμβουλίου, αλλά και στη δήλωση του Επιτρόπου Χάν, καθώ και στο τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα το Μάρτιο. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι το 2016 ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά για μας σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ένταξη τον Φεβρουάριο πέρυσι παρουσιάσαμε την υποψηφιότητά μας, υποβάλαμε την υποψηφιότητά μας ε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια ε, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων πήρε θέση και ζητήθηκε και η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 9 Δεκεμβρίου λάβαμε και ένα ερωτηματολόγιο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα λοιπόν με όλους τους δείκτες, το 2016 ήταν το έτος το πιο επιτυχές, αν θέλετε, για τη Βοσνία σε ό,τι αφορά τον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, το Συμβούλιο Υπουργών είναι ε, ένας κινητήρας, μια μηχανή για την ένταξη. Γι' αυτό το πετύχαμε μέσα σε λίγους μήνες, μέσα σε δύο χρόνια. Βεβαίως, για να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε τα δύο τελευταία χρόνια, αναγκαστικά να περιμένουμε νωρίτερα 7 χρόνια. Είχαμε υπογράψει μια συμφωνία συνεργασία το 2008. Σε μια εποχή που η Βοσνία και η Τζοκοβίνη ε, δεν είχε πολύ καλές σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες ε, των ε, Δυτικών Βαλκανίων, έξω από την Κροατία ε, βεβαίως υπήρξαν πολλά προβλήματα τα οποία μπορέσαμε όμως να ξεπεράσουμε. Γι' αυτό λοιπόν το 2016 είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας. Ήταν η ευρωπαϊκή χρονιά της Βοσνίας από τότε που ξεκίνησε η ενταξιακή διαδικασία. Το, το 2016 συνέχισε την εντατική εργασία της στο Υπουργικό Συμβούλιο της Βοσνίας, διότι γνωρίζουμε ότι αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που παρουσιάζει τις περισσότερες προκλήσεις και σε διοικητικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι με βάση όλες τις αυτές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε προετοιμασμένοι. Ε, έχουμε μια φιλοδοξία, την ίδια φιλοδοξία που αναφέρει ουσιαστικά η εντολή μας να λάβουμε δηλαδή ε, το καθεστώς της υποψήφιας χώρας έως το πρώτο τρίμηνο του ερχόμενου έτους. Είναι φιλόδοξος στόχος, αλλά είναι εφικτός, διότι βασίζεται σε ρεαλιστικά στοιχεία και βεβαίως πρέπει να δούμε και τα χαρακτηριστικά των χωρών που μας περιβάλλουν. Θα πρέπει να υπάρξει μια επαγγελματική και τεχνική προπαρασκευή για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερωτηματολόγιο τη Κομισιόν και θα χρειαστούμε και ένα μηχανισμό συντονισμού που να λειτουργεί εξαιρετικά. Θα ήθελα να πω ότι όλα τα όργανα που συμμετάσχουν στο συντονισμό είναι ενημερωμένα και πληρούμε όλες τις διοικητικές προϋποθέσεις και όλες τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο αυτόν και να απαντήσουμε στο ερωτηματολόγιο. Αυτή η πρώτη φάση, η απάντηση στο ερωτηματολόγιο έχει ολοκληρωθεί. Τώρα περιμένουμε, αναμένουμε συνεργασία σε όλα τα επίπεδα ε, στη Βοσνία Τζαγοβίνη. Όλοι μας βοήθησαν. Έχουμε 20.000 σελίδες απαντήσεις στο ρηματολόγιο. Είχαμε βέβαια πάνω από 3.000 ερωτήσεις. Ε, ολοκληρώσαμε λοιπόν με επιτυχία αυτή την περίπτωση και αυτή την φάση μάλλον και τώρα περνάμε στην επόμενη. Ε, έχουν δημιουργηθεί κάποιες ομάδες εργασίας ε, ε, στα πλαίσια της συντονιστικής ομάδας. Ε, εκεί θα γίνει μια τεχνική δουλειά που θα συνεισφέρει στην απάντηση στα ερωτήματα. Αυτή η διαδικασία θα αφορά 25.000 σελίδες απαντήσεων. Θα χρειαστούμε χρόνο βέβαια για να τη συντάξουμε, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το ολοκληρώσουμε εντός των επόμενων μηνών. Οι θεσμοί της χώρας μου θέλουν να επικεντρωθούν στην ποιότητα των απαντήσεων, όχι μόνο στην ταχύτητα με την οποία θα δοθούν. Εμείς ακολουθούμε τις ενδείξεις που μας ε, έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσουμε, ακολουθούμε τις οδηγίες της Κομισιόν δηλαδή, ελπίζουμε να ακολουθούμε τη διαδικασία αυτή των επόμενων μηνών και έτσι ε, στο πρώτο εξάμεινο του ερχόμενου έτους ελπίζουμε να μας χορηγηθεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. Κυρίες και κύριοι, η Βοσνία Ερζεγοβίνη κάνει ό,τι μπορεί για πλήσει τις προϋποθέσεις ε, της Συμφωνίας Σταθερότητας και Συνεργασίας. Έχουμε πολλές συναντήσεις με τον ίδιο στόχο. Ε, τον περασμένο μήνα είχαμε μια συνάντηση στο Σαράγεβο. Ε, το Συμβούλιο σταθεροποίηση και Σύνδεσης θα αρχίσει να λειτουργεί και στις Βρυξέλλες. Το να συνέρχεται εκεί. Σε ό,τι αφορά τώρα το κοινοβουλευτικό σκέλος μετά την πρώτη συνάντηση που έγινε στο Σαράγεβο το 2015, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική επιτροπή μας. Αυτή η κοινοβουλευτική επιτροπή εργάζεται Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η διάσταση κοινοβουλευτική της συμφωνίας έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Από όσο ξέρω, με βάση το που μου οι εκπρόσωποι αυτής της Επιτροπής, τα προβλήματα που παραμένουν θα επιληθούν ε, σύντομα, μετά από δύο χρόνια εργασίας. Έτσι λοιπόν, τα μέλη της Επιτροπής εδώ θέλουν να, να επενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να εγκριθεί αυτός ο κανονισμός. Το Συμβούλιο Υπουργών για να μπορέσει να φτάσει στις προτεραιότητες αυτές ε, που αναφέρουν στην έκθεση της Κομισιόν ε, έχει στρωθεί στη δουλειά. Έχουμε ένα δεσμευτικό έγγραφο το οποίο θα εφαρμόσουν οι θεσμοί της χώρας και στην περιοχή του Μπρίτσκο. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη εξακολουθεί να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται. Είναι ένα πακέτο κοινωνικονομικών αλλά και νομικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζεται από κοινού με το σχέδιο δράσης. Από τα 34 μέτρα τα οποία αφορούν δικές μας αρμοδιότητες, τα 18 έχουν ήδη εφαρμοστεί και 7 είναι εν εξελίξη. Πιστεύουμε λοιπόν αυτή η ατζέντα μεταρρυθμίσεων στην Βοσνία Τζεγοβίνη ό,τι αφορά το Συμβούλιο Υπουργών έχει επιτευχθεί σε ένα ποσοστό 53% έχει υλοποιηθεί. Ε, Βεβαίω μιλάμε μόνο για δύο χρόνια, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε για 80% αφού είναι μόνο δύο έτη. Τώρα, σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχουμε εγκρίνει τα μέτρα σε επίπεδο 40% και σε ό,τι αφορά τη σερβική δημοκρατία 50%. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η ατζέντα μεταρρυθμίσεων στην Βοσνία Ζεγοβίνη υλοποιείται από κινούμενο σχέδιο δράση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σε γενικέ γραμμέ για το σύνολο τη χώρα το ποσοστό υλοποίηση είναι του 50%, είναι 50%. Αυτό που θα θέλαμε να αναφέρουμε επίσης είναι το θέμα των δημοσίων μισθών, των μισθών στο δημόσιο μάλλον, να βελτιώσουμε ε, και το σύστημα φορολόγησης αλλά ε, και την αγοραστική δύναμη. Ε, έχουν, έχουμε αυξήσει τις δυνατότητες που έχουμε σε φορολογικό επίπεδο, σε επίπεδο ίσπραξης δηλαδή, ίσπραξη των ε, φόρων το 2016 είχαμε μια αύξηση 4% σε σχέση με το 2015 και φέτος έχουμε πάλι αύξηση 4%. Αυτή η ατζέντα μεταρρυθμίσεων έχει οδηγήσει στο να σταθεροποιήσουμε τα οικονομικά μας ε, καθώς ε, και ο δείκτης πιστοληπτικός, σύμφωνα με τη Moody's, το 2017 εξακολουθούμε να έχουμε θετική, θετικές τάσεις. Θα πρέπει βεβαίως να βελτιώσουμε και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε εδώ και δύο χρόνια και υπάρχουν αποτελέσματα. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ, του πραγματικού ΑΕΠ για το 2015 είναι στους 3%, το 2016 2,8% και οι προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας πριν από μερικές εβδομάδες αναφέρουν ότι φέτος θα είναι πάνω από 3,2% ο αριθμός ανέψυξης και πάνω από 4% του χρόνου. Η ανταγωνιστικότητα των βοσνιακών επιχειρήσεων επίσης βελτιώνεται. Αυξάνονται και οι εξαγωγές. Αυτό είναι ένας δείκτης ανάπτυξη νομίζω για τη χώρα μας. Το 2016 είχαμε αύξηση των εξαγωγών στις τάξη του 4%. Το 2016 επίσης είχαμε αύξηση των εξαγωγών και μείωση του ελλείμματος. Τα αποτελέσματα για φέτος θα είναι σίγουρα τα καλύτερα των τελευταίων 20 ετών. Αύξηση των εξαγωγών 13% ...40% σε πέδο σέφτα, αλλά και σε πέδο έχουμε αύξηση. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία οι εξαγωγές προς την Ευρώπη για τη Βοσνία είναι εξαιρετικά ε, σημαντικές. Επίσης αναπτύσσεται ο τουρισμός. Από το 2015 είχαμε αύξηση ε, της τάξης του 20%, πάνω από 20% και διανεκτερεύσεις. Το 2016 είχαμε αύξηση και των ε, των, των τουριστών αλλά και την εκπαιδεύσεων σε ξενοδοχεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια γενική τάση άυξησης ε, στον τουρισμό της τάξης του 25%. Σε κάποιους τομείς είμαστε, παίζουμε γενικό ρόλο στην περιοχή, στην ενέργεια, στην παραδοσιακή, παραδοσιακή, παραδοσιακή βιομηχανία. Είμαστε γνωστοί ε, ε στον τομέα της μεταλλουργίας, ε, της ε, ε, αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχουμε κάνει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις για την περίοδο 2017-2019, μεταρρυθμίσεις ε, διαστρωτικές που θα μας επιτρέψουν να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη, να υπάρξει σταθερότητα και να εφαρμοστούν και μέτρα ε, εξοικονόμησης. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας και σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς στην περιοχή και αυτό αποτυπώνεται ε, στις εξαγωγές μας που είναι εξαγωγές εξαιρετικά ποιοτικέ. Τέλος, τους τελευταίους 20 μήνες έχουν δημιουργηθεί πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. Έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στους πιο νέους, διότι η ενεργεία των νέων είναι το μεγαλύτερο μακροοικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Από αυτού λοιπόν ε, εργαζόμαστε. Οι σχέσει καλής γειτονίας τώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να εφαρμοστούν οι εξωτερικές, για να εφαρμοστεί η εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο με τις χώρες της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε δημιουργήσει πλαίσια συνεργασία όπως η διαδικασία του Βερολίνου ή οι έξι των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης το Μάρτιο φέτος στο Σαράγεβο είχα την τιμή ε, να υποδεχθώ μια σειρά από ηγέτες της περιοχής, ήταν και ο Πίτροπος Χάν, ήταν και εκπρόσωποι από την Ιταλία. Αυτή η συνάντηση ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Εν πάση περιπτώσει, η συνεργασία εξακολουθεί να είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα η οικονομική. Η οικονομική συνεργασία θα είναι και το θέμα που θα εξεταστεί στην επόμενη βαλκανική συνάντηση τους επόμενους μήνες. Τον Φεβρουάριο επίσης υπογράψαμε μια συμφωνία στον τομέα των μεταφορών που κάτι που συμβολικό είναι εξαιρετικά, συμβολικά είναι εξαιρετικά σημαντικό με τη συμμετοχή των διαφορών ηγετών των βαλκανικών χωρών. Μετά τη συνάντηση λοιπόν στην θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους ε, γείτονές μας ε, για να ολοκληρωθούν τα διάφορα προγράμματα τα οποία συμφωνήθηκαν στην Τεργέστη. Σε αυτήν τη συνάντηση ε, ελπίζω να οριστούν οι προσπάθειές μας στην Τεργέστη, να έχουμε την έγκριση κάποιων εγγράφων αλλά και των διαφόρων μέτρων που έχουμε εγκρίνει. Ελπίζουμε να υποστηρίξετε οικονομικά ε, τις, ε, τα project που έχουμε υποβάλει. Μεταξύ των project, project αυτών δεν υπήρχε κανένα βοσνιακό σχέδιο ε, πέρσι, διότι δεν ήταν έτοιμη τότε η πολιτική μας στον τομέα των μεταφορών. Τώρα όμως έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε εργαστεί σε ό,τι αφορά την υποδομή στον τομέα των μεταφορών, αλλά και σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό τομέα, Νομίζω ότι πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε και η χώρα μας να συμμετάσχει σε αυτή τη χρηματοδότηση. Επίσης έχουμε εγκρίνει μια στρατηγική περιβαλλοντική που περιλαμβάνει αυτά που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Νομίζω λοιπόν ότι το πακέτο μεταρρυθμίσεων μας ε, και σε αφορά διασυνδέσεις μεταφορών είναι κάτι το οποίο έχει στεφθεί από επιτυχία. Ελπίζω λοιπόν τα προγράμματα που έχουμε υποβάλει επτά προγράμματα στον τομέα των μεταφορών, στον τομέα του περιβάλλοντος, στον τομέα του πολιτισμού, ε, μεταξύ άλλων. Ε, ελπίζουμε λοιπόν να ληφθεί υπόψη η τεχνική ποιότητά τους ε, να εγκριθούν και να υποστηριχθούν στην Σύνοδο Κορυφής της Τεργές της. Αυτό θα ήταν και η καλύτερη, το καλύτερο κίνητρο για τη χώρα μας για να μπορέσει να συνεχίσει να επενδύει, να βελτιώνει το επίπεδο ζωής των συμπολιτών μας. Πέρα από την περιφερειακή συνεργασία, ενισχύσαμε και τις διμερείς σχέσεις με τις χώρες της περιοχής. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο, να ενισχύσουμε την περιφερειακή συνεργασία και να έχουμε μια πολιτική καλής γειτονία και συμφιλίωσης. Στο τέλος του 2015, στο Υπουργικό Συμβούλιο συναντήσαμε την κυβέρνηση της Σερβίας και φτάσαμε σε συμφωνία, κάποιες διμερείς συμφωνίες. Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο φέτος επισκεφθήκαμε την κυβέρνηση και της Σερβίας αλλά και του Μαυροβουνίου και στις 6 Ιουλίου θα οργανώσουμε μια κοινή συνάντηση του δικού μας Υπουργικού Συμβουλίου και της κυβέρνησης της Κροατίας στο Σαράγεβο. Στη συνέχεια υπάρχει το άρθρο 15 της Συμφωνίας Σύνδεσης ε, και Σταθεροποίησης. Βεβαίως και θα σεβαστούμε εμείς το άρθρο 15 και ε, έχουμε συνεργαστεί με το Μαυροβούνιο προς την κατεύθυνση αυτή αλλά και με τη Μακεδονία. Ε, έχουμε υπογράψει συμφωνία φέτος. Υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο των συγκεκριμένων σχέσεων ακόμα. η θέσπιση των οριστικών συνόρων. Εμείς συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας σε ό,τι αφορά τα σημεία διέλευσης μεταξύ Βοσνίας και Κροατίας και Βοσνίας και Σερβίας. Έχουμε εξαρτητικές πληροφορίες από αυτού, υπάρχει ένα σχέδιο δράσης για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία και με τις δύο χώρες σε ό,τι αφορά τα κοινά μας σύνορα. Στο περιθώριο της νότου Κορυφής της Βιέννης ε, φτάσαμε σε μια συμφωνία συνοριακή με το Μαυροβούνιο, το οποίο, η οποία εφαρμόζεται. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό για μας. Ελπίζουμε όλοι οι Ευρωπαίοι φίλοι μας να μας βοηθήσουν να επιληθεί οριστικά το θέμα αυτό των συνόρων. Κυρίε και κύριοι, η Βοσνία Ζεγοβίνη κάνει την το της ε, στα πλαίσια της συνεργασίας ε, για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ένωσης και υποστηρίζουμε την, την θέση της Ένωσης ε, και την πολιτική της. Θα βοηθήσουμε στην εφαρμογή στο μέτρο που βεβαίως των νοτοτήτων μας. Η Βοσνία, Ζεγοβίνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζονται πολλές κοινέ προκλήσεις. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να συνεισφέρουμε στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Υπήρου, στην πρόθεση της δημοκρατίας, της ειρήνης, του κράτους δικαίου σε όλο τον κόσμο. Φτάσαμε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενός πλαισίου συμμετοχής της Βοσνίας στις επιχειρήσεις, της, της διαχείρισης κρίσεων. Σε αυτή τη συμφωνία εμείς ε, απευθυνθήκαμε στην Υπατία εκπρόσωπο και στις ε, αρμόδιες αρχές του τομέα της ασφάλειας ε, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να συμμετάσχουμε σε αυτές τις αποστολές. Η Βοσνία Τζεγοβίνη είναι ένας εταίρος αξιόπιστος, ένας εταίρος αποφασισμένος με αποφασιστική δράση ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξίσουμε την ασφάλεια και ξέρουμε βεβαίω τις ευθύνες που υπάρχουν στον τομέα της ασφάλειας. Όταν η Βοσνία Ζεγοβίνη προείδρευσε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης μάλλον, ε, εγκρίθηκε ένα κείμενο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των ξένων μαχητών. Επίσης εγκρίναμε ένα πρωτόκολλο, ένα επιπλέον πρωτόκολλο, ήμασταν η έκτη χώρα που το επικύρωσε και τέθηκε σε ισχύ, σε ισχύ μάλλον την 1η Ιουλίου φέτος. Η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι η πρώτη χώρα της περιοχής που τροποποίησε το ποινικό δίκαιο για να τιμωρούνται οι ξένοι μαχητές που φεύγουν από τη Βοσνία και πάνε να πολεμήσουν στο εξωτερικό. Έχουμε και μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη το 2016 στη χώρα μας δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση ξένου μαχητή. Το 2016 δεν είχαμε επιστροφή ε, χιλιάδων μαχητών από τη Συρία, όπως μας έλεγαν κάποιοι. Ε, είναι 46. Οι 40 αυτή τη στιγμή διώκονται και οι άλλοι 6 περνούν από εξονοχιστικό έλεγχο από τις αρχές μας. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές, τις υπηρεσίες πληροφοριών μας και η τάση για το πρώτο εξάμεινο φέτος είναι η ίδια. Δηλαδή δεν υπάρχουν Βόσνοι υπήκοοι που να πηγαίνουν, ε, να φεύγουν, να πολεμήσουν στο εξωτερικό. Θα ήθελα επίσης να πω το εξή. Εμείς θα επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας κατά της τρομοκρατίας για να υπάρξει καλύτερη πρόληψη της βίας, της ριζοσπαστικοποίησης, του εξτρεμισμού. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε βέβαια και με άλλε χώρε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια πρόκληση. Συνεργαζόμαστε επίση για την αντιμετώπιση του ξυλίματο χρήματο και που, που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. Επίσης ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δυνατότητε και μηχανισμού για να μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα παράνομε δραστηριότητε με στόχο την τρομοκρατία. Και θα πρέπει βεβαίω έγκαιρα να μπορούμε να, παγώνουμε, να δεσμεύουμε τα όποια μέσα χρησιμοποιούνται προ την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει η Βοσνία να βγει από, το, από τη λίστα φάτουα. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης δεν είμαστε στις υπόλοιπες λίστες, ελπίζουμε να μας βγάλουν και αυτή τη λίστα. Πέρυσι στην Επιτροπή αυτή ξεκίνησε μία πρωτοβουλία για διάλογο και σε πιο χαμηλό επίπεδο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων για να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην περιοχή και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς συνεργασίας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι η Βοσνία Ριζεγοβίνη εκτιμούν ιδιαίτερα τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να βοηθήσει τη Βοσνία στην πορεία της προς την Ευρώπη. Αυτή η ομάδα φίλων ε, της Βοσνίας ε, υπάρχει εδώ και ένα χρόνο και αυτό είναι εξαιρετικά ε, ευχάριστο. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να υποστηρίζει τη χώρα μας και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει στο μέλλον. Θα έχουμε ε, κοινέ εκδηλώσει ε, που θα επικεντρωθούν σε πολιτικά αλλά και σε άλλα ζητήματα. Οπότε δεν είναι απαραίτητα πολιτικά τομεί ε, όπου η Βοσνία θα μπορεί να έχει μεγαλύτερη παρουσία όπω στον τομέα του πολιτισμού, διότι έχουμε ένα, μια κοινή, έχουμε μια πλούσια μάλλον συγνώμη πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά. Και σίγουρα ο πολιτισμό αυτό ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο για τη Βοσνία αλλά και την ευρύτερη περιοχή και για ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, υπάρχει ένα σχέδιο πολύ σημαντικό, το Μουσείο Αρσέιβικ, το οποίο αποτυπώνει την αλληλεγγύη ε, και στο οποίο συμμετέχουν διάφοροι καλλιτέχνες της χώρας μου. Τέλος, η αλλαγή του εκλογικού νόμου, της εκλογικής νομοθεσίας. Όλοι γνωρίζουμε στη Βοσνία ότι πρέπει να υπάρχει μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το κενό που υπάρχει ε, το κενό που υπάρχει μετά την απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων. Υπάρχουν δύο αποφάσεις. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, διότι εάν δεν εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις, θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα Αυτές οι αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου ζητούν αυτό το σύστημα των τριών εθνικοτήτων να μην εφαρμοστεί στις εκλογές, διότι αυτό οδηγεί σε διακρίσεις. Αν αυτή η απόφαση Σέιντιτ Φίντσι δεν εφαρμοστεί, ουσιαστικά αντιβαίνουμε τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις απαιτήσει του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, όπως, αυτά, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αποφάσεις του. Όλοι θέλουμε βεβαίως αυτός ο εκλογικός νόμος να αλλάξει. Είναι απαραίτητο να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του, του, δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του ΕΔΑΔ. Και αυτό πάει πέρα από την εθνική νομοθεσία της χώρας μου. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην γίνει σεβαστή αυτή η απόφαση. Όπω είπα, εμεί θα εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντα υπόψη τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και τις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Θα ήθελα τώρα ε, να ζητήσω από όλους τους φορείς να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους ε, για να μπορέσουμε να πετύχουμε όλες τις ε, προϋποθέσεις για να πετύχουμε το στόχο μας. Και το πιο σημαντικό σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων είναι να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Στην περίπτωση της Βοσνίας αυτό είναι θεμελιώδες, διότι εμείς δεσμευόμαστε να συμμετάσχουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, που είναι μια οικογένεια αξιών. Ειρήνη, δημοκρατία, κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα ε, και όλες τις λοιπές αξίες που περιλαμβάνονται στην πολιτική διεύρυνση. Εφαρμόσουμε την ατζέντα μεταρρυθμίσεων στη Βοσνία ε, και να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενσωματωθούμε, να ενταχθούμε στην Ευρώπη, να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τη Συμφωνία σύνδεση και Σταθεροποίησης, να βελτιώσουμε τη συνεργασία. Όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητες ε, για μας. Θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε αποφασισμένοι, το Υπουργικό Συμβούλιο της Βοσνίας είναι αποφασισμένο ε, για να συμμορφωθεί, να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα ε, προς την ευρωπαϊκή ένταξη προς όφελο των πολιτών της Βοσνίας και της Ζεκοβίνης. Οι πολίτες της χώρας μου Αναμένουμε ανυπομονησία αυτό το καθεστώς υποψήφια χώρας, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις. Ιδάλω ε, θα έχουμε σημαντικέ ε, ε και αυτό θα αυξήσει και τις επιφυλάξεις που υπάρχουν. Ελπίζω λοιπόν να μας υποστηρίξετε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι εξωτερική πολιτικής της ε, χώρας μου. Θέλω να επαναλάβω και εγώ με τη σειρά μου της, ε, στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου ε, όσον αφορά την ανάπτυξη των ε, δυνατοτήτων να καλωσορίσω μάλλον άλλη μια φορά τους βουλευτές της Βοσνίας Ερζεγωμένης, την πρώην Δημοκρατία της ε, της ε, Μακεδονίας, ε, τους εκπροσώπους του Μαυροβουνίου, της Μολδαβίας και όλων των υπόλοιπων χωρών. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Πρέντα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα εδώ σε αυτήν την Επιτροπή ένα χρόνο ε, αργότερα. Να σας ευχαριστήσω και για την πολύ επικοδομητική συνεδρίαση που κάνουμε στο Σαράγεβο πριν από καμιά δεκαριά μέρες, όπου μας υποδεχτήκατε τόσο ωραία εμένα και το συνάδελφο Πιτσούλα από την ε, Σοσιαλιστική Ομάδα. Το είπα στο Σαράγεβο, αλλά το λέω και ξανά εδώ, ότι έχετε την πλήρη μας υποστήριξη όσον αφορά τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την ε, πρόθεση της ολοκλήρωσης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα από όσα είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και σας συγχαίρω προσωπικά και πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μεταρρυθμιστές όπως εσείς. Να σας ενθαρρύνουμε να προχωρήσετε, να συνεχίσετε και για να αντισταθούμε σε ένα είδος αντίληψης που έχει κάπως ε, εμπεδοθεί, ότι δηλαδή ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων έχει ε, ε, καθυστερήσει. Πιστεύω αντίθετα ότι εσείς έχετε κάθε βούληση να προχωρήσετε σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και παράλληλα με τις απαντήσεις που δώσατε στα ερωτηματολόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ξέρω πως θέλετε και εσείς όπως και εμείς η Βοσνία Ζαγοβίνη σύντομα να αποκτήσει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. Αυτή λοιπόν η πολιτική ε, όθηση είναι πολύ σημαντική, όπως είναι σημαντική και η συνεργασία και αναζήτηση συμβιβαστικών ε, λύσεων. Και είχα μάλιστα τη δυνατότητα, με, αφού ε, με υποδεχτήκατε στο Σαράγεβο να μεταβώ στην Πάνια Λούκα όπου διαβίβασα αυτό το μήνυμα και στις επαφές μου με τον κύριο Ιγκουρ Σέναβα που είναι υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της χώρας με τους συναδέλφους της Ρεπούμπλικα Σέρσκα, τους εθνικούς βουλευτές και με τον πρόεδρο Ντόντιτς που του είπα, του εξήγησα ότι είναι μέρος της διαδικασίας, ότι δεν είναι ο μόνος, δεν μπορεί να είναι ένας ξεχωριστός ε, συνομιλητής, αλλά ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί στην διαδικασία αυτή και κυρίως στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής δράσης, δηλαδή στο να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο. Και είμαι ευτυχής που είναι σήμερα εδώ οι συνάδελφοι ε, των κοινοβουλίων, γιατί δυστυχώς έχουμε πρόβλημα ακριβώς με τους ε, βουλευτές συναδέλφους. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε προσπαθήσει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε το ICPC και δημοσία κάνω έκκληση στους συναδέλφους, ιδιαίτερα στον κύριο Τάντιτς, για να ξεπεραστεί να, να ξεπεραστούν τα εμπόδια που μας εμποδίζουν να έχουμε επαφές ε, φυσιολογικά όπως κάνουμε σε όλες τις άλλες χώρες. Από ό,τι κατάλαβα ο κ. Στάρης άλλαξε γνώμη. Ελπίζω ε, να έχει ήδη ξεπεραστεί λοιπόν το εμπόδιο αυτό και ότι θα μπορέσουμε να συναντιόμαστε τακτικά ώστε να ακούμε πρώτα απ' όλα τα όσα έχουν να μας πούν οι συνάδελφοι της Βοσνίας Ερζεκοπίνης για αυτή τη διαδικασία. Δεν θα λάβουμε εμείς αποφάσεις για τη χώρα σας, δεν θέλουμε καθόλου να σας αντικαταστήσουμε εμείς, να σας υποκαταστήσουμε, δεν θέλουμε παρά να έχουμε μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ κύριε Τάντιτζε που μπορέσατε να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια. Και έχω και μια ερώτηση για εσάς, αν κύριε Πρωθυπουργέ μου το επιτρέπετε. Για εσάς ποιο θα ήταν το ιδανικό σενάριο για το ερωτηματολόγιο, για τις απαντήσεις και τη γνώμη της Επιτροπής. Πότε θα είστε εσείς ικανοποιημένο να έχετε την απάντηση και πότε θα είναι υποψήφιο στην ολοκλήρωση, υποψήφιο μάλλον προς ολοκλήρωση η χώρα σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίτσουλα. predsjedavajući, ε, doista ja se radujem što smo danas ovdje ugostili gospodina Denisa. Ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερως που έχουμε τον κύριο Ντένις Σβίτζιτς μαζί μας ανάμεσα σήμερα. Ε, ε, είχαμε μία εβδομάδα μονάχα ανάμεσα στις ε, δύο ε, συναντήσεις. πρόσφατα στο, βρέθηκα στο Σαράγεφο και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογό μας. Αρχικά λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ τον επικεφαλής διότι μας παρουσιάσετε πολύ καλούς δείχτες για το έργο της κυβέρνησής σας κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι η Βοσνία Ριζεκοβίνη μπορεί να εργαστεί πολύ καλά και να ε, επιληθούν προβλήματα παρά τους ε, πολύπλοκους θεσμούς ε, και τις πολιτικές συνθήκες εν ώψη ε, αυτών ε, που θέλουν να επιταχύνουν την πρόοδο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, γνωρίζετε ότι έχετε φίλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι θέλουν να σας βοηθήσουν για να ξεπεράσετε τα εσωτερικά και εξωτερικά σας προβλήματα αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσετε και μια καλύτερη κατανόηση σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική της ευρωπαϊκής της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ε, ε, η αναφορά του 2014 και 2015 ε, επιβραδύθηκε όμως η κατάσταση το 2016. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω δύο πράγματα σχετικά με την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων που προβλέπετε να κάνετε στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Το πρώτο αφορά ένα φαινόμενο το οποίο ε, παρατηρείται σε αρκετές χώρες της ε, Βαλτικής αλλά και, της, ε, και των Βαλκανίων που αφορά την διαρροή εγκεφάλων από το πιο παραγωγικό κομμάτι του πληθυσμού και τις σοβαρές δημογραφικές, πολιτικές και οικονομικές συνέπειες από τη δεκαετία του 1990 λοιπόν πάνω από 23 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ε, φύγει από αυτές τις ε, περιοχές προς τη Δυτική Ευρώπη. Έχετε λοιπόν κάποιες προφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σχετικές ε, για την μεταπολεμική κατάσταση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Και ως επικεφαλής λοιπόν του Υπουργικού Συμβουλίου έχετε κάποια μέτρα υπόψη τα οποία θα μπορούσαν να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν αυτή την έξοδο ε, νέων ανθρώπων από τη χώρα σας ε, και επίσης ε, ποιος θα είναι η βάση αυτών των μεταρρυθμίσεων σε περίπτωση που φύγουν όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τον κοινωνικό διάλογο στη χώρα σας. Όλες οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους κοινωνικούς εταίρους ούτω ώστε να γίνεται μια σωστή αναδιανομή των βαρών των μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένας κοινό διάλογος των μέτρων που εφαρμόζει κυβέρνηση παρέμβασή ε, και ε, θα ήθελα δημοσίως ε, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την υποστήριξη και για το γεγονός ότι δύο χρόνια συνέχεια η διαδικασία για τη δημιουργία μιας κοινή κοινοβουλευτική επιτροπής για την σύνδεση συνεχίζεται, θα συνεχιστεί ούτω ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή. Σα ζητώ να είστε πιο σύντομοι για να μπορέσει να έχει το χρόνο να απαντήσει ο Πρωθυπουργό. Ευχαριστώ. Κύριος Ράντο. Ε, σας καλωθορίζουμε εδώ πέρα κύριε ε, ε, τα ε, μέλη του Κοινοβουλίου της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης, εξοχότατε κύριε Πρέσβη. Ευχαριστούμε πολύ που, μιλού, που μιλήσατε για ε, την κατάσταση και τις εξελίξεις της Βοστίας Ζεγοβίνης ε, στην έκθεση των τελευταίων μηνών αλλά ε, και για τα οικονομικά ζητήματα ε, σχετικά με την φορολογία για παράδειγμα. Παρά όλα αυτά όμως υπάρχουν πολλά τα οποία ακόμα ε, πρέπει να γίνουν. Το 58% των εισαγωγών καλύπτεται από εξαγωγές. Έτσι λοιπόν η Βοσνία Ερζεγοβίνη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί. Το ερώτημα μου τώρα προς εσάς αφορά τα ερωτηματολόγια και απαντώντας τα ερωτηματολόγια σίγουρα θα χρειαστείτε έναν συντονισμό ε, για τις δομές ε, της κυβέρνησης, ε, για, σε επίπεδο κυβέρνησης και οντοτήτων. Έτσι λοιπόν οι μηχανισμοί των οποίου, τους οποίους έχετε υιοθετήσει είναι οι πιο πολύπλοκοι μηχανισμοί συντονισμού που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής ε, προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τις απαντήσεις ε, για αυτά τα ερωτηματολόγια για την Βοσνία Ζεγοβίνη στο σύνολό της. Ε, χρησιμοποιείτε λοιπόν αυτό τον συντονιστικό μηχανισμό και πώς ακριβώς το κάνετε αυτό. Αυτή ήταν από τους βασικότερους όρους για την συνέχιση των θετικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και ταυτόχρονα αποτελούν και δείκτη σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ε, για ε, τον, ε, τη λειτουργία των συντονιστικών μηχανισμών και πώς θα εφαρμοστούν και σε άλλα στάδια των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. αναφέρατε μερικά ε, βήματα τα οποία θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχετε την πλήρη υποστήριξη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πρέντας χαίρομαι ιδιαίτερο στο ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών και όσο το δυνατόν γρηγορότερο όμως υπάρχει μία έλλειψη διαφάνειας ε, από την πλευρά των βοσνιακών αρχών σχετικά με το πώς ε, συμπεριλαμβάνεται το κοινοβούλιο και αυτό περιλαμβάνει βέβαια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακαδημαϊκούς και ούτω καθεξής. Και εφόσον συζητάμε περί διαφάνειας, η, ε, ε ευρωβουλευτές έστειλαν έγγραφο επιστολή στους θεσμούς αλλά και στο Συμβουλίο σχετικά ε, με το πώς ε, θα μπορούσε να σωθεί ε, ένας τηλεοπτικός σταθμός της χώρας σας και το μήνυμα από εμάς ήταν ότι η λήξη του BHRT ε, θα ήταν κάτι απαράδεκτο, θα ήταν η πρώτη χώρα χωρίς εθνική τηλεόραση. Τι λοιπόν σκέφτεστε για όλο αυτό, διότι δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση μέχρι στιγμής ε, και θέλουμε να ρωτήσουμε αν θα μπορούμε να προσδοκούμε σε μια απάντηση από εσάς. Κατανοούμε ότι χρειάζεται οικονομική ε, βοήθεια και φυσικά θα πρέπει να γίνει και μια ανάλυση του προβλήματος σχετικά με το πόσο σταθμό αυτό αυτός θα μπορέσει να συνεχιστεί στο ε, πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ε, ερώτησή μου. Τώρα όσον αφορά την καταπολέμηση της δημοκρατίας, ε, της ακρεοποίησης και τα λοιπά. μας δώσατε κάποιες πληροφορίες, όμως αναρωτιέμαι πώς συνεργάζεστε με, συνεργάζεται με άλλες χώρες της περιοχής, διότι αποτελεί ένα ζήτημα ασφάλειας Υπάρχει ένας φόβος στην περιοχή, έτσι λοιπόν πόσα δεδομένα ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών, τι μπορούμε να περιμένουμε από τη Βοσνία Ζεγοβίνη ε, στον τομέα της καταπολέμησης της ακροποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρωθυπουργός έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και για τις ευχές σας να γνωρίστηκαν οι προσπάθειές μας και η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα μας ε, στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Έχουμε ενισχύσει το κράτος δικαίου, έχουμε ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία και αυτό κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια. Εγώ μπορώ να πω με περηφάνεια ότι έχουμε επανέλθει στο δρόμο τον οποίο βρισκόμασταν εδώ και χρόνια και ελπίζουμε ότι θα μας φέρει προς την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αποχωρήσει λοιπόν η ολοκλήρωση και η συνεργασία με τις ε, και γειτονικέ χώρες. Να συνεχίσω λοιπόν να απαντήσω σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορώ. Ο κύριος Πρέντα που είναι και φίλος μου μίλησε για αυτό το ερωτηματολόγιο και για την δυναμική που ακολουθείτε με αυτό το ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι θεσμοί της ε, Σερβικής Δημοκρατίας έχουν αρχίσει να εισάγουν ε, τις απαντήσεις ε, σε αυτό το σύστημα το ενιαίο. Αν και έχουν χαθεί ήδη τέσσερις μήνες σχεδόν. Οπότε επιτέλους θα δώσουν μια κοινή απάντηση τους, τους επόμενους μήνες. Το σημαντικό είναι να μην γίνουν περισσότερες ερωτήσεις, αλλά να αρχίσει η αξιολόγηση της ποιότητας των απαντήσεων και στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους να λάβουμε θετική γνώμη και ότι τελικά θα μας ε, δοθεί το καθεστώς υποψηφίου. Θέλω να πω άλλη μια φορά ότι είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι, είμαστε δεσμευμένοι σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Για μας δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Είναι ο μόνος δρόμος τον οποίο εμείς θέλουμε να διανύσουμε. Ε, και γι' αυτό και εφαρμόζουμε όλες αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις που είναι πολύ οδυνηρές και δύσκολες. Ε, ε, πιστεύω πως αξίζουμε. Αξίζουμε το καθεστώς του υποψήφιας χώρας. Αξίζουμε να πάψει αυτό το μπλοκάρισμα που έχει κρατήσει εδώ και τόσα χρόνια. Και μάλιστα η Συμφωνία Σταθεροποίησης έχει υπογραφεί πριν από 8, σχεδόν 9 χρόνια. Και όλο αυτό το καιρό, όλο αυτό το διάστημα, εμείς, εκτός από από την ε, Κροατία, πέρα από την Κροατία, ήμασταν στην καλύτερη θέση. Δεν θέλουμε να πέσουμε θύματα περισσότερων ε, ε, άλλου παγώματος. Θέλουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να προχωρήσουμε στο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να τηρήσουμε τα όσα έχουμε υποσχεθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι επίσης πολύ σημαντικό να βασιζόμαστε σε έναν μοναδικό ενιαίο κανονισμό όσον αφορά αυτήν την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή η οποία θα ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Ακούσαμε τόσο είπε ο κ. Στάντιτς ε, αυτές τις δηλώσεις ε, ε, μετά από την τελευταία αυτή ε, συνεδρίαση. Είναι σημαντικά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Ανοίγεται ο, λοιπόν η πόρτα μετά από τα τελευταία ε, προβλήματα των δύο περασμένων ετών. Γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης πως ο κ. Στάντιτς ε, Βλέπω ότι γνέφηκε αυτός καταφατικά. Ναι, από ό,τι φαίνεται ναι. Τώρα, ερωτήσεις του κυρίου Πίτσουλα. Το θέμα των νέων η φυγή των εγκεφάλων είναι πρόβλημα για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και όχι μόνο να υπάρχουν πολλοί νέοι ε, που φεύγουν, αλλά φεύγουν γενικά νέοι από τις ε, χώρες, ε, από τα Δυτικά Βαλκάνια, γι' αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. στα προγράμματα ανάπτυξης και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης, κίνητρα για τους νέους, κυρίως για τους νέους και θέσεις κυρίως για τους νέους. Πιστεύω πως για να λυθεί αυτό το πρόβλημα χρειάζεται να υλοποιηθούν δύο προγράμματα, δηλαδή να ε, συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης. τελευταίους 11 ε, μήνες, 20 μήνες συγγνώμη, έχουμε δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στην πραγματική οικονομία. Πολλές από αυτές τις θέσεις είναι για τους νέους και χρειάζεται επίσης να μεταρρυθμιστεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ε, πιστεύω πως αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο σύντομα, ώστε να αναγνωρίζεται η ε, συμβολή της χώρας και φυσικά αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τους νέους είναι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και φυσικά όλα αυτά θα προχωρήσουν μέσω των ε, διαβουλεύσεων των ε, τοπικών ε, και αρχών κάθε περιφέρειας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης όπου λαμβάνονται νομοθετικά μέτρα ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματά τους στην απασχόληση και σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Και κάτι ακόμα, όπου όλοι συμφωνούμε, πρέπει να διατηρηθεί ένα επίπεδο ανεξαρτησίας πολιτικής και οικονομικής, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αντιπροσωπεύσουμε καταλήλως τους εργαζόμενους της χώρας μου. Άλλη ερώτηση του κυρίου Ράντος. η Επιτροπή Συντονισμού ε, υπάρχει και ε, σε όλους τους θεσμούς της ε, Βοσνίας της Στο πλαίσιο αυτού του μέσου συνεργασίας έχουμε δημιουργήσει 32 ομάδες εργασίας με πάνω από 1.500 μέλη που προέρχονται από όλα τα επίπεδα του διοικητικού μηχανισμού της Βοσνίας της Πρόκειται για πλήρη μέλη και για, για αναπληρωματικά μέλη που αντιπροσωπεύουν όλα τα θεσμικά όργανα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Επίσης αντιπροσωπεύονται εκεί και τα καντόνια και όπως βλέπουμε υπάρχει πλήρη συντονισμός για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε μια κοινή απάντηση ε, στα ερωτήματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερώτηση της κυρίας Φαγιών. Μιλήσατε για την ε, ραδιοτηλεόραση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και τις δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Εμείς από την πλευρά της κυβέρνησης ε, πιστεύουμε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι επαγγελματικού τύπου και ε, να παρουσιάζουν τις πληροφορίες ε, ε, προς τον λαό της Βοσνίας Ζεκοβίνης και να διαβιβάζουν τις επιτυχίες των διαφόρων διοικητικών αρχών, τοπικών και εθνικών. Θα πρέπει επίση να διατηρηθεί ο διεθνή χαρακτήρα τη Βοσνιακής ραδιοτηλεόρασης. Τώρα περιμένουμε πρόταση νομοσχεδίου που θα επιλύει το θέμα το, της βοσνιακής ραδιοτηλεόρασης. Και αυτό το σχέδιο νόμου τελικά Ελπίζουμε πως θα εγκριθεί εντός ολίγου και θα επιτρέψει την επίλυση του προβλήματος αυτού. Και όσον αφορά τη συνεργασία μας με άλλες ε, γειτονικέ χώρες για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό, έχουμε υπογράψει συμφωνία με την Europol που έχει μπλοκαριστεί για πολύ καιρό, αλλά τώρα ήδη έχει απεμπλακεί η κατάσταση και συνεργαζόμαστε στενά με τα όργανα της αστυνομίας καθώς και με τις μυστικές υπηρεσίες διαφόρων χωρών και μέσω της Europol και με την ε, ε, περιφέρειά μας, αλλά και με όλες τις χώρες του κόσμου, με τη ΣΥΠΑ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η τρομοκρατία είναι παγκόσμιος κίνδυνος, η παγκόσμια απειλή, από την οποία κανένας δεν μπορεί να προστατευτεί απολύτως, όμως μπορούμε να εργαστούμε προληπτικά και σε αυτό επικεντρωνόμαστε να διατηρήσουμε το στάτους ε, που έχουμε. Όπως ε, σας είπα, σε φέτος δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση τρομοκρατικής απόπειρας ή εξτρεμιστικής πράξης ή ε, πράξης ε, έλλειψης ανοχής ή κατά κάποιας εθνοτικής μειονότητας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και πρέπει να αλληλοβοηθούμαστε κατά κάθε είδους εξτρεμισμού και ριζοσπαστικοποίηση. Σας ευχαριστώ. Αντίο, και το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε καταφέρει Χάρη, ε, ελπίζουμε ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι, γιατί μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας συμφιλίωσης ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας ε, και για τη σημερινή σας πρόσκληση. Θέλω ακόμη μια φορά να επιβεβαιώσω ότι είμαστε προσιλωμένοι στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομική μας ανάπτυξη. Είμαστε υπέρ του κράτους δικαίου και υπέρ της περιφερικής συνεργασίας, ιδιαίτερα με τους γειτονές μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία αμοιβαία ε, συνεννόησης και συμφιλίωσης. Σας ευχαριστώ όλους για τα όσα έχετε κάνει ο καθένας με οργανωμένα και ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Ελπίζω πως και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να είμαστε ειλικρινεί εταίροι όπως ήμασταν μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Καλή τύχη. Bueno, continuamos, por favor. Συνεχίζουμε παρακαλώ ησυχία. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, οι πολιτικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Θα εξετάσουμε για δεύτερη φορά το σχέδιο έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας της Επιτροπής ΑΦΕΤ για τις πολιτικές σχέσεις με, την, με τον ΑΣΕΑΝ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ήταν 3 Μαΐου. Έχουν υποβληθεί 162 τροπολογίες συνολικά, 15 συμβαστικές τροπολογίες ε, που έχει προτείνει ο εισηγητής. Θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στον εισηγητή, τον κύριο Μπουτικόφερ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη αναφέρεται ότι ε, κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε σε συνολικά 15 ε, συμβαστικές ε, θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις για τον πολύ επικοδομητικό διάλογο και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, η οποία επίσης υποστήριξε το έργο μας, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για τη βοήθεια που μας έδωσε. Ε, όσον αφορά την ε, τροπολογία νούμερο 6, ε, παράγραφο 6, κατά λάθο και λυπάμαι για αυτό, η ε, γλώσσα έχει παραληφθεί από ε, την ε, συμβιβαστική, όμως έχουμε ε, συμφωνήσει στην συνάντηση των σκιωδών. Θα ήθελα λοιπόν να ενημερώσω όλους ότι σκοπεύω να συμπεριλάβω μια προφορική τρομολογία αύριο για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε αυτό ε, και η μία πρόταση ε, που θα πρότεινα να προσθέσουμε ε, ως προφορική τροπολογία στο τέλος της έκτης τροπολογίας έχει ως εξής υπογραμμίζουμε το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω εμπλοκή στην περιοχή και σε όλες τις διαδικασίες της ΑΣΕΑΝ. Θα ήταν μια παράβλεψη εάν δεν εκφράζαμε αυτή την βούληση και ε, δεν ε, υπήρχε καμία διαφωνία για αυτό το, ε, συγγνώμη για αυτό το πρόβλημα. Τώρα το δεύτερο σχόλιο το οποίο θα ήθελα να σας κάνω αφορά την παράγραφο 10 της ε, έκθεσης που προτείνει ε, να γιορτάσουμε ε, την φετινή επέτειο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΣΕΑΝ με ένα ε, πρόγραμμα ανταλλαγής το οποίο θα γίνει στο πλαίσιο της Προεδρίας της Σιγκαπούρης το 2018 με ενημέρωσαν από το Γενικό Γραμματέα της ΕΙΕΔ ότι η ΕΙΕΔ είναι διατεθειμένη να υποστηρίξει όλη αυτή τη διαδικασία μέσω, μέσω ε, το, του εργαλείου της εταιρική σχέσης, οπότε υπάρχει υποστήριξη και για αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα κύριο Στάνοκ δεν ζήτησα το λόγο, όμως χαίρομαι ιδιαίτερος που μου δίνετε ο λόγος. Είναι μια πάρα πολύ καλή αναφορά και χαίρομαι που ε, συμμετέχω ως ε, ε, Πολλοί προσπαθούν να συγκρίνουν την ΑΣΕΑΝ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πρόωρο, που είναι μια διαφορετική συλλογή κρατών όσον αφορά τον τρόπο διακυβέρνησης, τους πολιτισμούς, τις σχέσεις που έχουν και πιστεύω ότι στο μέλλον θα γίνει ε, μια εσωτερική αγορά με την οποία θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει ε, μια εμπορική σχέση. Όμως απέχουμε από μια τέτοια τελωνιακή ένωση, όμως ε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις που, ενισχυ... που ενθαρρύνουν τα κράτη ΑΣΕΑΝ να συνεργαστούν ούτως ώστε να ολοκληρωθούν περισσότερο στον τομέα του εμπορίου ε, και των οικονοποιών, αλλά όσον αφορά και την ε, συνεργασία των επιχειρήσεων. Ε, αυτή είναι μια λίστα επιθυμιών, ένα όρομα για το μέλλον και θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον κύριο Μπιτικόφα για το έργο του και εμείς θα υποστηρίξουμε όλες τις συμβιβαστικές. Ευχαριστώ, Σόλτς. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον γνωμοδότη για την έκθεσή του αλλά και την συνεργασία του που είχαμε αλλά και για τις συμβιβαστικές. Βλέπω ε, μια ε, σειρά ε, τροπολογιών και προτάσεων ε, για τον ε, τομέα αυτών. Η παραταξή μας το έχει σκεφτεί. Εμείς θα επιθυμούσαμε να ήμασταν πιο θαραλέοι όσον αφορά τις τροπολογίες και ιδιαιτέρως όσον αφορά την, τα ζητήματα της ενίσχυσης του διαλόγου για την κοινωνία των πολιτών Συνολικά λοιπόν ε, πιστεύω ότι ε, θα, με, όσον αφορά την ε, ψηφοφορία θα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη θέση όσον αφορά τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις αλλά και τη συνεργασία με τα κράτη ΑΣΕΑΝ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μίλερ. Πιστεύω ότι είναι μια καλή αναφορά ε, όσον αφορά την ε, συμβιβαστική ενέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαίρομαι που συμπεριλαμβάνεται αυτή. Με την άδειά σας ε, βλέπω ότι ο κύριος Πουσίνη είναι εδώ πέρα και θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι ότι χαιρετίζουμε τον πρώτο πολιτικό διάλογο που έγινε τον Οκτώβριο του 2015 και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν και άλλοι τέτοιοι πολιτικοί διάλογοι και θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί σημαντικό σε περίπτωση που ακολουθήσει ένας ακόμα τέτοιος πολιτικός ε, διάλογος ε, ε, στο πλαίσιο της 40ης επαιτίου των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πουσίνη θα μπορούσε να δώσει απάντηση πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η απάντηση του κυρίου Πουσίνη. Ε, με τα χαράς να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Έχουμε ε, προσπαθήσει επανειλημμένως ε, και πέρσι με την Προεδρία του Λάος να οργανώσουμε μια δεύτερη, ένα δεύτερο διάλογο, όμως εν τέλει ήταν αδύνατο για μια σειρά λόγων ε, ζητήσαμε λοιπόν από, τις, από την Προεδρία της, ε, των Φιλιππίνων ε, και εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή ούτως ώστε να οργανώσουμε τον δεύτερο διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ίσως να γίνει το Νοέμβριο. Εξετάζουμε αυτή τη στιγμή την ημερήσια διάταξη, τις ημερομηνίε, το πρόγραμμα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις πιθανές δυσκολίες που υπάρχουν υπάρχουν, όμως ε, πάντοτε έχουμε ξεκαθαρίσει προς τους ε, εταίρους μας και φίλους ε, στην ΑΣΕΑΝ ότι ο πολιτικός διάλογος τον οποίο οργανώσαμε το 2015 στις Βρυξέλλες δεν θα πρέπει να είναι μια και μοναδική πρωτοβουλία, όμως θα πρέπει να είναι ένα σύνθες χαρακτηριστικό των σχέσεών μας. Εργαζόμαστε λοιπόν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτόν τον δεύτερο διάλογο τον Νοέμβριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει σύντομα να επιβεβαιωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο αυτό. Αύριο ψηφίζουμε και το Σεπτέμβριο βεβαίως στην Ολομέλεια ξαναψηφοφορία. Πάμε στο επόμενο σημείο της εμείς διάταξης τώρα. Α, συγγνώμη, είχατε ζητήσει το λόγο για αυτό το σημείο. Εκτός μικροφώνιο, μιλήτρια όμως. Ναι, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Μιλάω εκ μέρους του κύριου David Μάρτιν για το σημείο αυτό, διότι δεν μπόρεσε να παραστεί. Αυτό που ο κύριος Μάρτιν θα ήθελε να πει είναι να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του και βεβαίως Χαιρόμαστε που καλύπτονται μια κλειδιά της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή καθώς και ε, το μέλλον της περιοχής αυτής. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΑΣΕΑΝ να συνεχίσουν και να βαθύνουν τις σχέσεις τους. Ο ΑΣΕΑΝ δεν είναι ο πιο σημαντικός εταίρος ε, εμπορικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά είναι μια περιοχή που από στρατηγική σημασίας είναι όλο και πιο σημαντική στο νέο, στη νέα τάξη πραγμάτων. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε πώς ασάν θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Στην Ασία ο ΑΖΕΑΝ έχει τη δυνατότητα να παίξει ένα ρόλο κλειδί για ζητήματα όπως η επίλυση διαφορών στην θάλασσα της Νοτιού Κίνας, καθώς και τα ζητήματα ε, αηφόρων άπτυξης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικά, ε, και μη συμβατική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να προσφέρει προς τον ΑΖΕΑΝ ως υπάρχον μοντέλο ε, περιφερειακής ολοκλήρωσης έχει προωθήσει την ειρηνική συνεργασία, την ανάπτυξη των εξεκρατών μελών εδώ και δεκαετίες. Έχει δημιουργήσει ε, δυνατότητες θεσμικές, έχει δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Μπορούμε λοιπόν να του βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε του ασιάτε εταίρου μα προ την κατεύθυνση αυτή. τη τροπολογία μα. η, η ομάδα μα έχει πολλέ πολλές τροπολογίε, πολλέ από αυτέ έχουν σωματωθεί στο συμβαστικό κείμενο. Όμω θέλουμε να ευχαριστήσουμε του κοιόδη εισηγητέ που εργάστηκαν για να ληφθούν υπόψη όλε αυτέ οι απόψει. Κάτι το οποίο David, ε, για το οποίο ο David ανησυχεί είναι ότι πρέπει να είμαστε φυλακτικοί στις σχέσεις της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ΑΖΕΑΝ, διότι αυτή τη στιγμή εξετάζεται η εμπορική συμφωνία και το θέμα ε, των εμπορικών συμφωνιών, ε, συμφωνιών ελευθέρων αλλαγών μεταξύ των δύο περιφερειών. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ και όχι σε ιστορικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λέει ο Ντέιβιντ. Ευχαριστούμε όλους του συναδέλφου για τη συνεργασία. Η ομάδα S&D θα υπερψηφίσει με χαρά αύριο ε, αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα με τη δεύτερη εξέταση του σχέδιου έκθεσης ε, των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολιτικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία. Είναι η δική μας ε, έκθεση που θα ψηφιστεί. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, Πρόεδρε, ήθελα μόνο να αντιδράσω με μία φράση στο σχόλιο της συναδέλφου σχετικά με τη σχέση μεταξύ πολιτικών και εμπορικών ζητημάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο της Επιτροπής ΙΝΤΕ, το είδα μαζί του, έτσι ώστε η διατύπωση σε αυτή την έκθεση ε, να μην τύχει αντίδραση στην Επιτροπή ΙΝΤΑ. Ευχαριστώ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν ξέρω να δίνω το λόγο σε κανένα για το θέμα αυτό. Η έγκριση λοιπόν προβλέπεται στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου αμέσω πριν τη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία που θα λάβει χώρα τέλο του έτου στο Νέο Δελχή. 194 τροπολογίε έχουν υποβληθεί, 17 συμβαστικέ τροπολογίες έχει υποβάλει ο εισηγητή. Θα δώσω το λόγο θύσαμε αμέσως στον εισηγητή, ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα ε, να καλωσορίσω, να χαιρετήσω τις συζητήσεις που είχαμε με τις άλλες ε, με του άλλου συγκητέ και όλου συγκητέ για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία. Από αυτέ τι ε, διαπραγματεύσει προέκυψε ότι μεγάλο μέρο ε, τη Επιτροπή μα επιθυμεί να ενισχυθούν οι σχέσει μεταξύ αυτών των δύο δημοκρατιών και ελπίζω η ευρενή ψηφοφορία να το επιβεβαιώσει αυτό. Ε, είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα δώσει μια όθηση στην Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία που θα λάβει χώρα το φθινόπωρο. Στα πλαίσια αυτή τη βούληση προσέγγισης και των συμβαστικών προτάσεων που διαπραγματευθήκαμε, μια σειρά από συγκεκριμένε προτάσει έχουν υποβληθεί για την σωστή εφαρμογή. Είπαμε στην αρχική έκθεση ότι πρέπει να αναπτύξουμε σαφείς ιδέες, σαφείς απόψεις για την Ινδία και για την γύρω περιοχή που παίζει να... έχει έναν περιθωριακό ρόλο στην στρατική μας ε, την παγκόσμια η Ατζέντα 2020 Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκού Ινδίας που εγκρίθηκε στι τελευταίε νοδοκορυφή θα πρέπει να υλοποιηθεί γρήγορα και σοβαρά. Επίση, θεωρούμε ότι διαπραγματεύσει για μια συμφωνία δευτερών συναλλαγών θα πρέπει να επανεκκινήσουν έτσι ώστε να, ολοκληρώσουν, να αναπληρωθούν και να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα ε, και οικονομικά και ε, κοινωνικά και για τις δύο πλευρές. Επίση, οι συμβαστικέ προτάσει αναφέρονται στι μεγάλε δυνατότητε συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών Συνδία σε επίπεδο εξωτερική πολιτική, μια και έχουμε τι ίδιε προκλήσει να αντιμετωπίσουμε σε μεγάλο βαθμό. Ε, η ασφάλεια, έλλειψη ε, σεβασμού στο διεθνέ δίκαιο, εξτρεμισμό, ε, ε, παράνομη μετανάστευση, ε, ριζοσπαστικοποίηση, ένα ε, σε βάθο ένας σε διάλογος μεταξύ των δύο αυτών εταίρων και μια συζήτηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των εντάσεων και των σειράξεων στην κύριο περιοχή αλλά και σε διεθνέ επίπεδο θα ήταν κατά τη γνώμη μα εξαιρετικά σκόπιμο. Προ την ίδια κατεύθυνση ένας ε, ενισχυμένο συντονισμό σε επίπεδο θέσεων Ηνωμένων Εθνών στα Ηνωμένα Έθνη, όποτε αυτό είναι εφικτό, και μια δέσμευση υπέρ του σεβασμού του διεθνού δικαίου και από τι δύο πλευρέ θα έκανε ότι αυτή η εταιρική σχέση θα ήταν εγγύηση της εφαρμογής των κοινών μας αξιών σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον μια σειρά από ε, παρεμφερή ζητήματα αναφέρονται και στο αρχικό κείμενο αλλά και σε πολλές τροπολογίες που έχουν υποβάλει συνάδελφοι. Και αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία. Παραδείγματο χάρη, ασφάλεια στη θάλασσα, ιδιαίτερα ε, δράση κατά του, της πειρατείας στον Ειδικό ωκεανό. Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν εδώ να αναπτύξουν κοινέ πρακτικές. Το θέμα της εταιρικής σχέσης στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ενέργειας. Ε, εκεί χρειάζεται ενίσχυση ε, της εταιρικής σχέσης που δεν θα είναι μόνο υπέρ του περιβάλλοντος και της οικονομίας των δύο πλευρών αλλά θα δώσει και μια όθηση στη διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτών. Ένα άλλο τομέα που έχουν εντοπίσει πολλοί συνάδελφοι που έχουν προβάσει σχετικέ τροπολογίε είναι αυτό των ανταλλαγών προσωπικού ε, μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο επαγγελματιών σε μια σειρά αποτομής, σε επίπεδο φοιτητών, επιστημόνων, σε, πολιτιστικό επίπεδο. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ Ευρωπαίων και Ινδών. Ένα άλλο άξονα συνεργασία που χρήζει περαιτέρω προσοχή είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών, είτε μιλάμε για την ελεύθερη έκφραση, είτε μιλάμε για την ε, ελεύθερη άσκηση θρησκευτικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να βρούμε περισσότερου τρόπου για να προσπίσουμε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Να λοιπόν κάποια ζητήματα από τα οποία συμφωνήσαμε με του σχεδόν συγγητέ, Θέλω να του ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ στο ότι εάν θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα το οποίο θα ακουστεί και στα όργανα αλλά και στον νέο Δελχή, δεν πρέπει να το πνίξουμε μέσα σε λεπτομέρειες ε, που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία ή μέσα σε αντιφάσεις. Να επικεντρωθούμε λοιπόν στα κεντρικά, να τονίσουμε δηλαδή τη βούλησή μας της προσέγγισης, να εντοπίσουμε κάποιους τομείς δράσης όπου η συνεργασία μας μπορεί να έχει μια προσθέμενη αξία και βεβαίως σε συστάσεις ό,τι αφορά την εφαρμογή της συνεργασίας αυτής στους τομείς αυτούς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γκίλ. Η κυρία Γκίλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ επίσης ε, τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση και για την επικοδομητική του συνεργασία. Νομίζω πως αυτό το εκτιμούν όλοι οι σκιώδεις ε, της έκθεσης αυτής. Ήταν ε, πια καιρός και ήταν καλή ευκαιρία για μας για να εστιάσουμε τις, τις ε, σχέσεις Ένωσης και Ινδίας και έχουμε εντοπίσει το μίσο που μπορεί να υπάρξει δυναμικό για βελτίωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί πολλές ε, παγκόσμιες πολιτικές αλλαγές συμβαίνουν ιδιαίτερα σε σχέση με τις ΗΠΑ και την απομονωτική της ε, στάση. Και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία έχουν κοινά συμφέροντα επί των οποίων μπορεί να βασιστεί στενή συνεργασία και ο Κρίστιαν ήδη τα περιέγραψε πολλά από αυτά, αλλά ίσως να προσθέσω κι εγώ κάτι και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε ώστε να χειριστούμε τις κλιματικές αλλαγές και να εξασφαλίσουμε παγκόσμια δέσμευση στην ατζέντα του Παρισιού και έχουμε ένα σημαντικό σύμμαχο με την Ινδία. Διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας ε, στον Ειδικό κενό αλλά επίσης θα μπορούσε να είναι η Ινδία σύμμαχος στην ε, νότια και στην θάλασσα ε, της Κίνας, αλλά ένας τομέας τον οποίο δεν έχουμε εξετάσει αρκετά εις βάθος, αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης και επίσης έχουμε και πολλά κοινά συμφέροντα όσον αφορά την ενίσχυση της ε, ε, διαδικτυακής ασφάλειας η προτεραιότητα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο είναι οι ε, θέσει εργασίας και ανάπτυξη. Αλλά η συζήτηση και ο διάλογος με την Ινδία καθώς και η σύσφυξη των εμπορικών δεσμών θα μπορούσε να μας βοηθήσει και σε άλλους τομείς. Και μιλώντας για το εμπόριο είναι πολύ λυπηρό που δεν υπάρχει καμία πρόοδο στι διαπραγματεύσει για την FTA. Δεν είναι κάτι το οποίο τώρα θέλουμε να σκεφτούμε, αλλά 10 χρόνια τώρα έχουν περάσει και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ανάγκη να ενδυναμωθεί και πάλι αυτή η προσπάθεια. Αυτή η συμφωνία είναι σημαντική γιατί οι FTAs εκτιμάται ότι διπλασιάζουν τη, θα διπλασιάσει μάλλον τις εξαγωγές της Ένωσης προς την Ινδία, αλλά θα στείλει και ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα όσον αφορά την ευρωπαϊκή ισχύ και την παγκόσμια μας θέση μετά από το Brexit. Εμένα με θαρρύνει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες ε, κάποια ανοίγματα στη συζήτηση FTA στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Μόντι στην Γερμανία, την Ισπανία και την Φεργαλία και ίσως να αυτή να είναι μια καλή ευκαιρία για μας εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και για την Κομισιόν να προσπαθήσουμε να βασιστούμε σε, αυτή, σε αυτά τα καλά μηνύματα και ενδείξεις. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Προβλέπετε διεθνή επαφή τον Οκτώβριο στο Δελχή και γι' αυτό είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η επικοδομητική ε, προσέγγιση. Ως κοιόδης λοιπόν καλωσορίζω το γεγονός ότι έχουμε εξασφαλίσει διάφορες ε, τροπολογίες κλειδιά στις συμβιβαστικές και σε ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτό όσον αφορά το FTA, τη ε, κλιματικές αλλαγές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω πως η έκθεση έχει βρει σωστή ισορροπία. Παρακαλώ, με συγχωρείτε διακόπτη πρόεδρε, να ολοκληρώσετε. Είναι σημαντικό να έχουμε μια προσεκτική και ισορροπημένη έκθεση. Έχουμε και την παρουσίαση μιας μελέτης για την ενέργεια, γι' αυτό και παρακαλώ να είστε λίγο πιο περιορισμένοι στα λόγια σας. Ευχαριστώ. Τάνο. Θα είμαι σύντομο. Ε, θυμάμαι το 1999, ε, ήμασταν τότε με την κυρία Γκίλ ε, και είχαμε ιδρύσει τότε τον Σύλλογο Φίλη τη Ινδία. τότε λοιπόν ε, είχαμε προεδρεύσει την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ινδία. Η Ινδία είναι μεγαλύτερη δημοκρατία της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 του πλανήτη. Ε, θα, ο πληθυσμός της προβλέπεται να ξεπεράσει της ε, Κίνας. Έχει έναν μεγάλο ε, πολιτισμό. Έχουμε πολλούς, πολλούς τομείς κοινή συνεργασίας όπως είναι οι κλιματικές αλλαγέ, ο η παγκόσμια τρομοκρατία καθώς επίσης και η διατήρηση του παγκόσμιου εμπορίου καθότι η Ινδία είναι χώρα μέλος των BRIC και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα θα έχουμε ε, διαπραγματεύσεις ε, για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας. Υπάρχει μεγάλος πληθυσμός διασποράς από την Ινδία στα κράτη-μέλα και ιδιαίτερος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια το Brexit τα αλλάζει όλα αυτά, όμως κάτι το οποίο δεν συνειδητοποιούν πολλοί είναι ότι υπάρχουν δύο πρωθυπουργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ειδική καταγωγή. Ο πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Κώστα, ο οποίος είναι η καταγωγής, αλλά και ο νέος πρωθυπουργός της Ιρλανδίας ε, είναι Ινδικής καταγωγής. Ε, είναι, υπάρχουν ε, ισχυροί δεσμοί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν και της Ινδίας. Ο κύριος Μπούκνερ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Έχω όμως κάποια σχόλια όσον αφορά την συμβιβαστική 7 αναφέρατε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όμως ε, δεν αποδέχεστε την τροπολογία 100 η οποία αναφέρεται ε, στην αποθήκευση ε, ρυζιού και σιτηρών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την διατροφή ε, του πληθυσμού σε περίπτωση που πληγεί από τυφώνες. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεδομένων των συζητήσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για αυτό το θέμα ε, θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την ε, θέση της Ινδίας σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, το δεύτερο τώρα αφορά την πιο ισχυρή διατύπωση για τα εσωτερικά προβλήματα ιδιαιτέρως για τον θρησκευτικό εξτρεμισμό, για τις κάστες για την ε, θέση των δικαιωμάτων, ένα πράγμα το οποίο όμως ε, δεν ε, καταλαβαίνω αφορά τα, γεν, τα φάρμακα, τα γενώσιμα φάρμακα, όμως αυτό, αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα ήθελα να συμπεριληφθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Βερόνικα από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Παρακαλώ, εν συντομία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή αλλά και τους σκιώδες ε, για αυτήν την έκθεση. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για αυτό. Το ε, βρίσκω σημαντικό το γεγονός ότι το πλαίσιο, το περιεχόμενο της συγκεκριμένη έκθεσης ε, αναφέρεται σε ζητήματα συνεργασίας. Επιθυμούμε να επεξεργαστούμε ζητήματα τα οποία αφορούν την ολοκλήρωση των δυνατοτήτων των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να υπάρχει μια στρατηγική αξιολόγηση αυτών των σχέσεων την επόμενη χρονιά και προσδοκούμε την σύνδον, τη σύνοδο ε, το φθινόπωρο που θα ακολουθήσει αυτήν του 2016 καθώς επίσης και την Ατζέντα 2020 που θέσαμε σε αυτό το πλαίσιο και επίσης θα θέλαμε να ε, συνεχίσουμε να χτίσουμε πάνω στις δράσεις που ξεκίνησαν Επίσης, κάποιοι από τους διαλόγους που επικεντρωνόμαστε αφαιρώνουν την ε, την ασφάλεια στη θέση, θάλασσα. Ε, οι κλιματικές αλλαγές επίσης είναι κάποια από τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν διότι ε, υπάρχει μεγάλη ε, ανασφάλεια όσον αφορά τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ε, και επιθυμούμε να υπάρχουν συνεργασίες ε, σε όλο τον πλανήτη και ιδιαίτερα με μεγάλες δημοκρατίες όπως είναι η Ινδία. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική έχουμε κοινέ προκλήσεις, αναφέρεται μερικές από αυτές, υπάρχουν και πολλές ακόμα, μπορούμε να εργαστούμε και πάνω σε αυτό και επίσης θα πρέπει να υπάρξουν επαφές μεταξύ των ανθρώπων όπως είναι για παράδειγμα στο πλαίσιο του Erasmus Plus όπου έχει υπάρξει μια ε, ικανοποίηση ε, όπου έχει υπάρξει μια μεγάλη αύξηση τα τελευταία ε, χρόνια και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Αλλά και η επιστήμη είναι ένας τομέας που μπορούμε να συνεργαστούμε. Επιθυμούμε έναν διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα συνεχίσουμε να πιέσουμε πάνω σε αυτό την Ινδία. Όπως προανέφερα θα γίνει μια σύνοδος στο φθινόπωρο και πιστεύω ότι η συγκεκριμένη έκθεση θα συνεχίσει να ε, προσθέτει στις σκέψεις μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Ευχαριστώ την κυρία Κόντι. Αύριο ψηφίζουμε και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο παρουσίαση της μελέτης για την ενέργεια. Σας θυμίζω ότι πρόκειται για συνάντηση κλεισμένων των θυρών. Μόνο δηλαδή οι βουλευτές και το προσωπικό των πολιτικών ομάδων και ε, οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να αποχωρήσουν.